Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Καλημέρα σας. Ε, σήμερα είναι κάπως δύσκολη ημέρα. Πάντα οι πέμπτες είναι δύσκολες περίπλοκες για τους ευρωβουλευτές. Πάντως θα ήθελα να καλωσορίσω την Ομίγυρη και να κηρύξω την έναρξη με μικρή καθυστέρηση της συνεδρίασής μας, αυτής της έκτακτης συνεδρίας της Επιτροπής Γεωργίας, της 7ης Μαρτίου. Να στήσω συγγνώμη εκ μέρους του Πρόεδρου μας, του κυρίου Σεκέσκη, που δυστυχώς κολλείεται, δεν βρίσκεται καν στις Βρυξέλλες σήμερα το πρωί και μου ζήτησε να τον αναπληρώσω. Έτσι και θα κάνω. Έχουμε σήμερα το πρωί δύο πολύ σημαντικές παρουσιάσεις. Καταρχήν να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Φαντάζομαι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσω γιατί δεν έχω ανακοινώσεις. Με το σημείο 3, το πρώτο συστικό σημείο της ημερήσιας διάταξης, ε, με την πρώτη παρουσίαση της πρωινή μα συνεδρίασης που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε εκπροσώπους ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Γάλακτος που θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμα υπευθυνότητα αγορών που εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Γερμανική Ένωση Γαλακτοπαραγωγών. Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα ειδικό πρόγραμμα για το γαλακτοκομικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση κινδύνου ανισορροπίας της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων. Για το τελευταίο καιρό, μετά την κατάργηση των γαλακτοκομικών ποσοστών, είχαμε πρόβλημα ανισορροπίας στην αγορά και για να αποφύγουμε στο μέλλον τέτοιες ισορροπίες, έχουμε αυτό το πρόγραμμα υπευθυνότητε αγορών που ενεργοποιείται σε περίπτωση κρίσης στην αγορά γάλακτος. Χρησιμοποιείται ένας δείκτης ε, αγοράς για τον υπολογισμό της σταθερότητας και ένας συνδυασμό παρακολούθησης και ανταπόκριση στην αγορά θα μας επιτρέψει να προλάβουμε κάποιες κρίσεις, να αναγνωρίσουμε τον επικείμενο χαρακτήρα μιας κρίσης. Αυτό είναι το όνειρο του κάθε γεωργού, να προλάβει την κρίση και να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις για να την αποτρέψει. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν πρόταση. Και θα δώσω πρώτα το λόγο στους παρακαθημένους. Να καλωσορίσω καταρχήν τον κύριο Έρβιν Σόψες, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Γάλακτος και τρία από τα μέλη του Συμβουλίου αυτού, τον Ιωάννης Φάλερ, τον Μπόρις Γκοντούιν, ε, δεν ξέρω αν είναι και ο τρίτος εκπρόσωπος, ο κύριος Κάρταν Πόλσεν, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Γάλακτος. Καλώς ήρθατε λοιπόν και θα δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Σόπιες για 10 λεπτά για να μας κάνει την παρουσίαση αυτού του ενδιαφέροντος προγράμματος για την υπευθυνότητα των αγορών. Καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που βρίσκομαι εδώ και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνετε να σας μιλήσουμε εδώ πέρα Είμαστε τέσσερις εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Γάλακτος και είμαστε και οι τέσσερις γαλακτοπαραγωγοί στις χώρες μας και να σας πω ότι ε, έχω τρομάξει κάπως από τον αριθμό ευρωβουλευτών που βρίσκονται εδώ. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι αρκετά ενδιαφέρον ο τομέας του γάλακτος και αν είναι αυτή η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και της εμπλοκής των Ευρωβουλευτών ε, πρέπει να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε για το πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η Ευρώπη στο μέλλον. Λοιπόν, οι παρατηρήσεις μου ως αγρότης ε, και ω ε, πολίτης. Λοιπόν, για το θέμα τώρα, ποιο είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γαλακτος. Ε, σε αυτό εκπροσωπούνται 21 οργανώσεις γαλακτοπαραγωγών 16 χώρες εκπροσωπούνται από το Βέλγιο, Κροατία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετωνία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Ελβετία. Και νομίζω ότι είμαστε, θα έλεγα, ένας οργανισμός με αρκετή κινητοποίηση και ποιος είναι ο στόχος μας, η φιλοσοφία μας. Κοιτάξτε, για εμάς ε, το σημαντικότερο είναι εμείς ε, οι αγρότες να λαμβάνουμε μια τιμή που θα καλύπτει το κόστος της ε, παραγωγής αλλά και να είναι ένα δίκαιο εισόδημα για τους παραγωγούς γιατί το γάλα είναι ένα από τα πιο αξιόλογα προϊόντα που υπάρχουν. Κανένας άνθρωπος, κανένα ανθρώπινο όν δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε γάλα. Ξεκινάμε από παιδιά και από τα μοσχάρια ξεκινάει αυτή η υπόθεση. Κανένα παιδάκι, κανένα μωρό δεν μεγαλώνει με κοκακόλα. Ε, το πρώτο το οποίο τρώει είναι το γάλα. Πρόκειται λοιπόν για ένα, πολύ, ένα προϊόν υψηλής ε, διατροφικής αξίας και πίσω από κάθε λίτρο γάλα που παράγουμε βρίσκεται μια γελάδα. Αλλά και ένας αγρότης, ένας άνθρωπος και μια οικογένεια. Πίσω από κάθε λίτρο γάλα που παράγουμε υπάρχει μια επιχείρηση μια ιστορία. Νομίζω, θυμόμαστε όλοι, μετά τον πόλεμο, πόσο σημαντικό ήταν το να υπάρχουν αγρότες που θα θρέψουν τους πολίτες. αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η υπόθεση, γιατί οι γονείς μα, οι παππούδες μα έθρεψαν την Ευρώπη και οποιοδήποτε λέει σήμερα ότι οι αγρότες δεν τα βγάζουν ε, πέρα σήμερα και άμα δεν τα βγάζουν πέρα να σταματήσουν για να κάνουν καμιά άλλη δουλειά ε, δεν αντιλαμβάνονται γιατί δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε γιατί ακριβώς αυτή η ιστορία που υπάρχει ε, υπάρχει στα αγροκτήματά μας και όλοι οι γαλακτοπαραγωγοί είμαστε περήφανοι για τη δουλειά μας περήφανοι για τα αγροκτήματά μας και για το προϊόν το οποίο είναι πολύ υψηλής ποιότητας και παράγουμε για τους πολίτες. Και γεγονό είναι ότι έχουμε κρίσεις και σήμερα βρισκόμαστε σε κρίση. Από το 2008-2009 είμαστε σε κρίση. Ξεκίνησε το 2009 η μεγάλη κρίση του γάλακτος. Όταν οργανώσαμε τη μεγάλη απεργία τότε που ρίχναμε τα γάλατα στους ε, δρόμους όλες αυτές οι διαδηλώσεις ε, φτάσαμε ε, να έρθουμε και εδώ πέρα και ρίχναμε το γάλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω, ίσως πρέπει να το ξανακάνουμε, όπως μας ακούσετε. Αλλά για εμάς είναι σημαντικό σήμερα να είμαστε σε διάλογο με τους ευρωβουλευτές, με τους ε, πολίτες και το σημαντικότερο είναι πρώτα απ' όλα να εμποδίσουμε τις κρίσεις για να μην υπάρχουν καν και αυτήν την ε, στιγμή εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε κρίση για εμάς, ε, για την Ομοσπονδία. Είναι σημαντικό απόλυτα να υπάρχει μια βιώσιμη γεωργία για όλους τους ε, γεωργούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε μια παραγωγή γάλακτος σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης και για να διατηρηθεί αυτό χρειάζονται τιμές που θα καλύπτουν το κόστος και να δώσουν έτσι και στη νέα γενιά την ευκαιρία να κρατήσουν αυτά τα αγροκτήματα όπως κάναμε και εμείς. Τα πήραμε από τους πατεράδες μας, τους παππούδες μας και θέλουμε να διατηρηθούν σε μια σωστή κατάσταση, να τα δώσουμε σε μια σωστή κατάσταση στην επόμενη γενιά. Πώς έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Πολλοί θεωρούν ότι η κατάσταση είναι καλή. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπετε πως υπολογίσαμε σε 6 ευρωπαϊκές χώρες το κόστος παραγωγής και αυτή τη στιγμή κατά μέσο όρο στην Ευρώπη το κόστος είναι 43 cent. Η τιμή αυτή τη στιγμή είναι 35 cent όμως. Άρα εξακολουθούμε να χάνουμε 10 λεπτά του ευρώ σε κάθε λίτρο για να μπορέσουμε να καλύψουμε το κόστος. Γιατί λοιπόν ε, τα καταφέρνουμε να επιζούμε. Με τα 35 αυτά σεντ πληρώνουμε τις ζωοτροφές, ε, τις περισσότερες πιστώσεις μας, ε, τα δάνεια, αλλά κρατάμε τα αγροκτήματα γιατί οι αγρότες δεν πληρώνονται μισθό. Υπάρχουν γονείς, παππούδες, γείτονες, συγγενείς που πάντα ε, εργάζονται χωρίς ε, να πληρώνονται στα αγροκτήματα. Και ειδικά αυτό για έναν νέο που θέλει να αναλάβει το αγρόκτημα και ξέρει ήδη ότι δεν μπορεί να πληρώσει ένα μισθό. Είναι η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω, ξέρετε, τα νούμερα. Εάν δούμε πόσες χιλιάδες αγρότες, χιλιάδες οικογένειες που έζησαν από την Γεωργία έφυγαν τα τελευταία χρόνια, τα παράτησαν. Πόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας χάσαμε, πρέπει να ανησυχούμε πάρα πολύ για το ότι στο μέλλον δεν θα υπάρχουν πια αγρότες να αναλάβουν το επάγγελμα. Θα πάμε σε μια βιομηχανική γεωργία όπου η παραγωγή θα είναι στα χέρια μεγάλων εταιριών και κεφαλαιακών εταιριών. Να δούμε λοιπόν μια μικρή αναδρομή. Η Κομισιόν εισήγαγε το μέτρο αυτό, το εθελοντικό το 2016 και νομίζω ότι το μέτρο αυτό, το πρόγραμμα ε, ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Εάν δούμε πόσοι γεωργοί συμμετείχαν σε όλες τις χώρες και βλέπουμε την εξέλιξη της ε, τιμής ε, του γάλακτος το 2016 τον Ιούλιο ήταν 25 σεντ και ένα χρόνο μετά ήταν 34 σεντ και ξανά 25 λεπτά ήταν η τιμή του 2016 που έπαιρνε ο αγρότης ε, φαντάζεστε πως ήταν τα πράγματα τι από κεφαλαιοποίηση υπήρχε. Και ακριβώς ειδικά στις χώρες που λέγανε ότι δεν ε, θα λάβουν μέρος οι αγρότες, ειδικά σε αυτές τις χώρες, Γερμανία, Ολλανδία, Αγγλία, Ιρλανδία, υπήρχε τεράστια συμμετοχή. Καταφέραμε να ε, έχουμε σχεδόν ε, ένα 3 εκατομμύριο λίτρα γάλακτος που βγήκε από την αγορά. Α, το μεγάλο λάθος το 2016 ήταν ότι ενεργοποιήθηκε πολύ αργά αυτό το πρόγραμμα. Πολύ αργά. Πρώτα ε, δόθηκαν 500 εκατομμύρια ευρώ σε επιδότηση στους ε, αγρότες και λέγαμε ότι έτσι θα βοηθήσουμε τους αγρότες. Στους αγρότες δεν έφτασαν όμως αυτά λεφτά, έφτασαν 100 ή 1000 ευρώ. Η Κομισιόν μετά αγόρασε 400.000 τόνους και αποθήκευσε 400.000 τόνους σκόνη γάλακτος και νομίζω ότι και στο μέλλον θα πρέπει να αντιδράσουμε πάρα πολύ νωρίτερα. Τα πούλησε μετά αυτή τη σκόνη σε 1600 ευρώ τον, με τον τόνο. Μετά 1200 ευρώ το τόνο και είχαν λεφτά χώρια το κόστος αποθήκευσης. Αυτό δείχνει ότι τα μέτρα αυτά της κρίσης είναι πλέον πεπαλαιωμένα και δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Το πρόγραμμα ευθύνης της αγοράς. Λοιπόν, έχουμε ακριβώς αυτό το παρατηρητήριο για την ε, τιμή του γάλακτος. Δεν έχει νόημα όμως να παρατηρούμε την τιμή του γάλακτος. Πρέπει το παρατηρητήριο αυτό να γίνει κεντρική δομή όπου δεν θα παρατηρεί μόνο το γάλα, αλλά θα δρά όταν υπάρχει κρίση. Το πρόγραμμα αυτό, το πρόγραμμα ευθύνης της αγοράς θα πρέπει να εδρεωθεί στην νέα ΚΑΠ. Ως πρώτο σημείο θα πρέπει στο μέλλον να έχουμε έναν δίκτυ. Έναν δίκτυο ο οποίος θα λειτουργεί ως μπούσουλας για το πότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός της κρίσης. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιηθεί για να ενεργοποιεί το παρατηρητήριο τον μηχανισμό κρίσης για να μην υπάρχει καν κρίση όσον αφορά τον σχηματισμό αυτού του δίκτυ, εντάξει μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά αυτό το οποίο είναι απολύτως σημαντικό είναι η πλήρης κάλυψη του κόστους για τους αγρότες. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον Μπόρις, ε, ο οποίος ε, είναι υπεύθυνος για το πρόγραμμα αυτό και θα σας το εξηγήσει στα στοιχεία του. Μάλιστα, ευχαριστώ. Μια στιγμή, μια στιγμούλα. Θα ήθελα απλώς να πω, όχι για να δικαιολογήσω τους συναδέλφους λόγω της μικρής προσέλευσης, αλλά βρισκόμαστε προς το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας και συμπίπτουν πολλές συνεδριάσεις, γι' αυτό απουσιάζουν πολύ. Πάντως σας διαβεβαιώ ότι είχαμε πολύ άριθμες συζητήσεις για το γαλακτοκομικό τομέα και όλες οι πολιτικές ομάδες εκδήλωσαν ζωηρό ενδιαφέρον για το γάλα. Δεν θέλω να δημιουργήσετε εσφαλμένε εντυπώσεις λόγω της μικρής προσέλευσης, να την εκλάβετε ως αδιαφορία για το γαλακτοκομικό τομέα. Δεν το λέω αυτό για να δικαιολογήσω τους απόντες, αλλά συμπίπτει η σημερινή μας συνεδρίαση με τη συνεδρίαση άλλων επιτροπών και έχουν και άλλες υποχρεώσεις οι ευρωβουλευτές. Εν πάση περιπτώσει, ο συνάδελφός σας τώρα μπορεί να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε το λόγο. Λέγομαι Μπόρις Βοντρουά. Είμαι γαλακτοπαραγωγός στη Γαλλία, στην ανατολική πλευρά της Γαλλίας. Είμαι 3,5 χρόνια εδώ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γάλακτος και θα σας παρουσιάσω τις διάφορες φάσεις ε, του προγράμματος υπευθυνότητα αγορών και πώς ε, ε, ενεργοποιείται το σύστημα. Όπως είπε ο συνάδελφος, το να συνεχίζουμε να παράγουμε γάλα χωρί ε, ρυθμιστικό μηχανισμό είναι αυτοκτονικό και για του παραγωγού, αλλά και για του καταναλωτέ και για το περιβάλλον. Οπότε έχουμε κάτι να πούμε εδώ, έχουμε κάποιο λόγο. Και για να επανέλθω στο πρόγραμμα αυτό υπευθυνότητα αγορών. Καλύτερη πρόληψη παλά η θεραπεία. Οπότε η πρώτη προειδοποίηση, ο πρώτος συναγερμός είναι η μείωση ε, κατά 7,5% του δίκτυ από το 100. Ε, στόχος είναι να αποφύγουμε οποιαδήποτε πιθανή επικείμενη κρίση. Τι κάνουμε λοιπόν στο παρατηρητήριο αγοράς γάλακτος. Το παρατηρητήριο αγοράς γάλακτος ε, μας είπε ίσως ε, να κάνουμε αυτοκατανάλωση αντί για παράδοση γάλακτος. Να το χρησιμοποιήσουμε για την εκτροφή των μοσχαριών ή να βοηθήσουμε τους βιομηχάνους να κάνουν ιδιωτική αποθεματοποίηση, μικρής κλίμακος, μέχρι κάποια όρια βέβαια. Κατόπιν θα πρέπει να κρατήσουμε ένα υψηλό επίπεδο επαγρύπνησης μέχρι ότου επανέλθουμε στο δίκτυο 100. Καλύψουμε δηλαδή αυτή τη μείωση. Αυτά για την πρώτη φάση. Αν τώρα ο δείκτης πέσει κατά 15% από το 100, σημαίνει ότι ήδη μπαίνουμε στην κρίση. Οπότε το πρόγραμμα Επιθυνότητας Αγορών, το PRM, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο μηχανισμός του θα κινητοποιηθεί πανευρωπαϊκά. Οπότε ε, ορίζουμε και κάποια περίοδο αναφοράς και ε, τις ποσότητες ε, ε, που έχουν παραχθεί τις βλέπουμε για ένα χρόνο πριν την περίοδο και λέμε ότι θα πρέπει οι νέες ποσότητες να ξεπεράσουν αυτές τις, ποιο... τις ποσότητες αναφοράς. Επίσης, προβλέπεται και ένα πριμ. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί στα τέλη του 2016 είχαμε τους δύο τελευταίους μήνες του 2016 μία ρύθμιση που προτάθηκε με την καταβολή κάποιες πρημοδότησης. Και το σύστημα λειτουργήσε, γιατί ακόμη και χώρες όπως η Ιρλανδία, που ήταν ε, έτοιμες να ε, παράγουν με πολύ χαμηλό κόστος, δέχτηκαν αυτή την πρημοδότηση, αυτή τη μικρή ενίσχυση για να μειώσουν την παραγωγή τους. Και μας εθάρρυνε πολύ και μας ικανοποίησε αυτό το παράδειγμα γιατί μας έδωσε την ελπίδα ότι το πρόγραμμα υπευθυνότητας αγορών μπορεί να λειτουργήσει στην αγορά. Οπότε τίθενται ανώτατα όρια παραγωγής για τη συγκεκριμένη περίοδο σε όλες τις κτηνοτροφικές ομάδες. Και επίσης από το πρώτο κιλό υπερβάλλουσας ποσότητας επιβάλλονται πρόστιμα στους γαλακτοπαραγωγούς. Με, τη βάση, με βάση την αρχή ο Ριπένο πληρώνει. Αυτός που παράγει περισσότερο χρεώνεται για να μην πληγούν αυτοί που μείωσαν τις ποσότητες τους. Οπότε όσοι υπερβαίνουν την ποσότητα καταβάλουν πρόστιμο. Και στην τρίτη φάση, αφόσον ε, έχουν ενεργοποιηθεί βέβαια οι δύο προηγούμενες, δεν χρειάζεται καν να φτάσουμε στην τρίτη φάση. Βέβαια τώρα βρισκόμαστε στην τρίτη φάση, έχουμε πέσει κάτω από το 25% του κόστους παραγωγής. Οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργοποιήσουμε το τρίτο σκέλος του προγράμματος, δηλαδή υποχρεωτική πια μείωση της ποσότητας, ανελαίητα. Δεν δίνουμε τίποτα στους ε, παραγωγούς και τους υποχρεώνουμε να μειώσουν τις ποσότητες, ενώ στη δεύτερη φάση ήταν εθελοντική η μείωση της παραγωγής. Αυτά. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Θέλει κανείς άλλο το λόγο από το Συμβούλιο Γάλακτος, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γάλακτος τα συμπεράσματα, τα συμπεράσματα. Α, θα το κάνετε ντουέτο εδώ. Ωραία. Σύντομα όμως, για να έχετε το χρόνο μετά τη συζήτηση να δευτερολογήσετε. Να πω κάποιο συμπέρασμα. Απευθύνουμε έκκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εσείς είστε η ελίτ ε, των αιρετών ε, της Ευρώπης. Εσείς είστε οι αιρετοί που μας εκπροσωπούν ε, και δεν είστε υπάλληλοι όπως αυτοί οι οποίοι εργάζονται στην Κομισιόν. Αυτό ελπίζουμε ότι θα μας στήριξετε. Δεν θέλουμε επιδοτήσεις ε, πλέον στο μέλλον. Θέλουμε να μπορούμε να ζούμε από την παραγωγή μας. Τα παλαιά μέσα ε, πλέον δεν λειτουργούν. Έχει φτάσει η στιγμή να έχουμε ε, νέα μέσα. Έχουμε μέλλον τι θα γίνει με το Brexit αν πάει στραβά τι θα γίνει εάν σταματήσουν πάλι εξαγωγές ε, προς την Κίνα με κάποιο σκάνδαλο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν χρειαζόμαστε αυτό το πρόγραμμα. Δεν θέλουμε πλέον αποθήκευση στο μέλλον και θεωρώ ότι τώρα είναι η στιγμή να εισαχθεί αυτό το πρόγραμμα. Και τέλος θα ήθελα να πω γνωρίζω ότι ε, μιλάτε αυτή τη στιγμή για την Αφρικα Task Force και θα ήθελα να σα πω ότι είμαστε ε, απολύτως ε, κατά αυτών των φτηνών εξαγωγών αυτού του dumping ε, προς την Αφρική. 9 και 10 θα κάνουμε μια εκδήλωση μαζί με τους Αφρικανούς συναδέλφους μας, με τους αγρότες από την Μπουρκίνα Φάσο, Μαλή, Τσάντ, Μαυριτανία, Νίγηρα, για να σταματήσει η υπερπαραγωγή και το dumping προς την Αφρική. Σας ευχαριστώ που μας δώσατε τον λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Πολύ καλά συμπεράσματα. Περνάμε τώρα στη συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους που τον ζήτησα. Τρία λεπτά το πολύ παρακαλώ Πολυτέλεια είναι το τρίλεπτο. σύνηθω. έχουμε πολύ λιγότερο χρόνο. Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για ένα λεπτό μόνο. Τώρα έχουμε τρία ολόκληρα λεπτά. κυρία Σρέιερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω κάτι πρώτα απ' όλα στον Πρόεδρο της Επιτροπής εδώ των Γαλακτοπαραγών. Εγώ είμαι από μια οικογένεια, όλα μου τα αδέρφια μου ε, και τα νύψια μου ασχολούνται με την ε, κτηνοτροφία. Το ένα κομμάτι είναι στη δικιά σας οργάνωση και ένα άλλο κομμάτι της οικογένειας είναι στην άλλη οργάνωση και δίνει γάλα στην Καμπίνα και στους άλλους ε, συνεταιρισμούς. Λοιπόν, αυτό είναι γεγονός ε, ότι δεν συμφωνείτε ως γαλακτοπαραγωγή. Μπορείτε να μας ασκείτε κριτική, αλλά πρέπει να δείτε λίγο και τα δικά σας. Το είπε και η πρόεδρος. Ε, δηλαδή να υπάρχει και λίγος σεβασμός ε, για τους ε, εκπροσώπους που βρίσκονται εδώ πέρα. Εμείς ερχόμαστε σε σας έτσι το, το ξέρετε. Εγώ έχω κάθε διάθεση να σας ακούσω. Πάω και στην ε, σχετική οργάνωση που σας ε, ανέφερα. Λοιπόν, μιλήσατε και για την ε, κρίση. Έχουμε ακούσει και άλλους συναδέλφους σας Λοιπόν, δεν θα εξακολουθήσω, δεν θα εξαντλήσω τώρα τα τρία λεπτά. Λοιπόν, κοιτάξτε, έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές με την υπόθεση του γάλακτος και φροντίσαμε ακριβώς να ε, έχετε την ε, δίκαιη τιμή που θα έπρεπε να έχετε. Αλλά ξέρετε, δεν ε, οφείλεται σε εμάς το θέμα, είναι η εφαρμογή της οδηγίας. Τώρα, και έρχεστε και μου λέτε ότι δεν χρειαζόμαστε τη στήριξη του εισοδήματο. Μπορώ να σας πω, στην οικογένειά μου δεν συμφωνεί κανείς ε, με σας, ε, γιατί έχουν αυτή την επιδότηση για τα 200-300 εκτάρια. Έχουν επενδύσει πάρα πολλά λεφτά, αλλά δεν φτάνουν πράγματι αυτά για να υπάρξει κάποια καινοτομία. Οπότε, αυτό το οποίο θέλω να σας ρωτήσω. Εμείς εδώ πέρα είμαστε του ΕΛΚ. Καλό είναι να σκεφτούμε όλοι μαζί για κάποιες λύσεις σε αυτήν την κρίση. Αλλά κοιτάξτε, σας λέω την αλήθεια. Τα δύο τρίτα των ε, γαλακτοπαραγών στην Ολλανδία που γνωρίζω δεν συμφωνούν μαζί σας με αυτά τα οποία είπατε. Εντάξει, μπορείτε να κατηγορείτε τους ε, πολιτικούς, αλλά Μπορώ να μιλήσω και στα γερμανικά, αν θέλετε μαζί σα. δεν είναι πρόβλημα. Πώ μπορούμε να έχουμε κάποιε ιδέε για να έχει μέλλον η τομέα του γάλακτο. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ. Τρία λεπτά ακριβώ. Μπράβο σα. Έχετε φοβερή αίσθηση του χρόνου. Ο κύριο Ραπέ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που είναι παρόντες σήμερα. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Χαιρόμαστε που ήρθατε σε μας, που θίξατε τα προβλήματα και που προσφέρετε κάποιες λύσεις. Πρέπει να σας πω ότι πολύ συχνά έχουμε συζητήσει το πρόβλημα σε κάποιες χώρες ο γαλακτοκομικός τομέας είναι πιο σημαντικός από τις άλλες. Αλλά ο τομέας αυτός είναι πραγματικά σημαντικός για την επιβίωση του γεωργικού τομέα, της αγροτικής κοινότητας. Αυτοί που εργάζονται στο γαλακτοκομικό τομέα εργάζονται πολύ σκληρά. Από το ξημέρωμα μέχρι το βράδυ. Δεν έχουν διακοπές και η ζωή τους είναι πραγματικά δύσκολη. Επίσης, να πούμε ότι το 2015 έγιναν κάποιες προτάσεις. Προτάσεις για τη διακοπή του συστήματος ποσοστώσεων. Να θεσπιστούν ε, κανόνες, να δοθούν κίνητρα. Αυτό ίσως να βοηθήσει να διατηρηθεί ο τομέας. Ταυτόχρονα πρέπει να παραδεχτούμε ότι σε κάποια κράτη-μέλη επιδεινούται η κατάσταση. Και αν δεν κάνουμε τίποτα, τελικά θα φύγει ο κόσμος από τον τομέα, όπως γίνεται στη χώρα μου, στη Λιθουανία όπου μειώνεται ο αριθμό εκείνων που ασχολούνται με τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Και στο τέλος δεν θα έχουμε αρκετούς αγρότες και δεν θα μπορέσουμε γρήγορα να αποκαταστήσουμε τον τομέα. Χρειάζεται κάποια χρόνια μέχρι ότου να αρχίσει να, γίνει, να παράγει γάλα μια γελάδα. Πρέπει να σκεφτούμε και αυτή την πτυχή. ανησυχώ όπως και εσείς για αυτό που είπατε, για το εισόδημα των ε, γεωργών και τις δαπάνες. Αναφερθήκατε στα 10 cents διαφορά. Η κατάσταση είναι πραγματικά σοβαρή. Ε, σε κάποια κράτη-μέλη είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση από αυτήν που περιγράψατε. η μέση τιμής, η τιμή αγορά είναι 35 cents το κιλό. Σε κάποια άλλα κράτη-μέλη πάνε 40. Σε κάποια κράτη-μέλη μπορεί να είναι 27 και 28 ακόμα. Τα συστήματα πληρωμών διαφέρουν και αυτά ανάλογα με τα κράτη-μέλη. Κάπου οι πληρωμές είναι ψηλότερες, κάπου αλλού είναι χαμηλότερες. Ε, υπάρχουν κάποιες προτάσεις για τη δίκαιη ε, αμοιβή είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι η τιμή είναι το σημαντικότερο στοιχείο. Πρέπει να σκεφτούμε το πώς θα διαχειριστούμε την τιμολογική πολιτική στο γαλακτοκομικό τομέα. Αν πετύχουμε εκεί καλά αποτελέσματα θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά άλλα προβλήματα. Συμφωνώ με αυτό που είπατε. Η κυρία Μαγκίνης και άλλοι συνάδελφοι εργάστηκαν σκληρά για να πετύχουν ένα σύστημα δικαιότερης αμοιβή για τους παραγωγούς για τους μεταποιητές, για τους... Ε, Τελειώνεται κύριε Ροπέ. Ε, πιστεύω ότι το ΔΕΚ αποφάσισε ότι η κοινή αγροτική πολιτική ε, είναι πιο σημαντική από την ανταγωνιστική πολιτική, για την πολιτική ανταγωνισμού. Θα πρέπει να επιλύσουμε λοιπόν το πρόβλημα της τιμολόγησης. Ευχαριστώ κύριο Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε να πω στον πρώτο ομιλητή ότι θεωρώ ότι τα σχόλιά του είναι πολύ ε, σχετικά, πολύ σωστά παρατήρηση για τον αριθμό των μελών που είναι παρόντα. Να σας πω σαφώς, ίσως ο αριθμός των μελών να είναι μικρός, αλλά είμαστε καλοί και μπορούμε εύκολα να εκπροσωπήσουμε τη Γεωργία. Δεν χρειαζόμαστε όλη την Επιτροπή να είναι παρούσα. Διότι κάποιοι έρχονται εδώ μόνο και μόνο κάνουν ανακοινώσει στον τύπο. Εμείς είμαστε εδώ να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, απειλήσατε να σκορπίσετε γάλα στο κοινοβούλιο. Θυμάμαι, βρωμή ο τόπο για εβδομάδε. Μην το ξανακάνετε. Δεν σα βοηθά να κάνετε κάτι τέτοιο και δεν θα κερδίσετε φίλου αν το κάνετε αυτό. Αυτή είναι η Αν αυτή είναι η νοοτροπία σα, σα λυπάμαι. Διότι δεν ωφελείτε με αυτόν τον τρόπο τον τομέα σα, αν έτσι θα συμπεριφερθείτε στο μέλλον. Ένα πρόβλημα έχω από αυτά που άκουσα γιατί είναι πιο σημαντική αυτή που η γαλακτοκομία από αυτού που καλλιεργούν βόλιο, έχουν ζώα, βόλιο κρέα, χείριο κρέα κλπ. Γιατί είναι πιο σημαντική. Όλοι είναι εκεί, όλοι δουλεύουν, αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα ίδια προβλήματα. Λοιπόν, τελικά ε, θα καταστραφεί όλη η Ευρώπη και τα κοπάδια εάν αποτύχει ο τομέα. Είναι ένα από τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίσουμε στο Κοινοβούλιο. Έχω, έχω δει πολλέ κρίσει στο γαλακτοκομικό τομέα και ξέρετε σωστά, πολλά σωστά είπατε, πάρα πολλά. Όλοι ανησυχούν όταν συμβαίνει μια κρίση και διαμαρτύρονται και μόλις φύγει η κρίση όλοι τη λησμονούν. επιστρέφουν και παράγουν περισσότερο γάλα και αυτό κάνει αυτή τη στιγμή ο γαλακτοκομικός τομέας και οδεύει προς άλλη μια κρίση και τίποτα δεν έγινε μετά την τελευταία κρίση. Πρέπει να ενισχύσουμε το παρατηρητήριο τη αγορά. Έχετε δίκιο, πρέπει να το κάνουμε αυτό. Θα πρέπει να θεσπίσουμε νομοθεσία του στο πρόγραμμα να νομικά δεσμευτικό για όλα τα κράτη-μέλη. Πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά και τίποτα. Δεν έχει γίνει μέχρι την επόμενη κρίση. Και τότε όλοι θα κατηγορούν όλου του άλλου. Και κανεί δεν θα επομιστεί τι ευθύνε του. Εδώ έγκυται το πρόβλημα και η κρίση. από όταν εξαφανιστεί η κρίση, συνεχίζεται η ίδια συμπεριφορά. Την περασμένη φορά λέγαμε θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε εκείνο. Τι έγινε, τίποτα. Κάποια πράγματα έγιναν, αλλά κάποια πράγματα έπρεπε να γίνουν ή ξεκίνησαν και έμειναν ημιτελεί. Συμφωνώ μαζί σα, υποστηρίζω και η Επιτροπή θα σα υποστηρίξει, πιστεύω. Δεν είναι προ όφελο τη γεωργία. Δεν είναι προ όφελο του γεωργού συνεχώ να έχουμε τέτοιε διακυμάνσει. Τίποτα δεν είναι καλύτερο από ένα αμετάβλητο εισόδημα. Σταθερό εισόδημα. Και αν κάποιος θέλει να πάρει δάνειο, όπως ένας νέος που πρέπει να δανειστεί από τις τράπεζες και να έχει σταθερό εισόδημα για 5-10 χρόνια, είναι κάτι πολύ καλύτερο από κάποιον που θα βγάλει κέρδη μια χρονιά και θα έχει ε, απώλειες και ζημιά την επόμενη χρονιά. Αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε. Ε, και αυτή θα είναι η πρόκληση. Και άλλη μεγάλη πρόκληση για μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω μεγαλύτερη δυσκολία διότι οι γεωργοί μου θα αντιμετωπίσουν και το Brexit. Και για λίγο θα είναι καλά, σε καλή θέση. Ναι, ναι, το ξέρω, θα το πω, θα το πω. Και πιθανότατα θα είναι καλά μια χαρά, διότι έχουν πρόσβαση στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι 60% αυτάρκης όσον αφορά τα τρόφιμα που ζητούν. Αυτό για σύντομο διάστημα, μέχρι ότου η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου διαπραγματευτεί συμφωνίες με την Νότια Αμερική, με τις ΗΠΑ και όλους τους άλλους. Όλες αυτές είναι λύσεις βραχυπρόθεσμες. Βραχυπρόθεσμες δεν είναι καλές. Χρειάζεται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός που θα εφαρμοστεί και θα ελεγχθεί παντού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη που μακρηγόρησα. Το κυρία Χόιμπουχ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Ομοσπονδία Μωρίς Ιωάννης γνωριζόμαστε εδώ και χρόνια και πάντα εκτιμώ το ότι οι Ευρωπαίοι γαλακτοπαραγωγοί εντάξει μπορεί να είχαν κάποιες απο, ε, αποφάσεις οι οποίες δεν ήταν πάντα προς το συμφέρον μας γιατί και εγώ είμαι γαλακτοπαραγωγός πάντα έκαναν την προσπάθεια να βρουν ε, και να προτείνουν μια λύση εντός ε, του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Αυτή λοιπόν είναι μια πρόταση την οποία πρέπει να σκεφτούμε. Γιατί τα είπε και ο κύριος ε, Νίκολσον, πρέπει να εισαχθεί ένας αυτοματισμός ο οποίος θα κινητοποιείται όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτές οι αλλαγές στην αγορά. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας αυτοματισμός ο οποίος ακριβώς θα προλαμβάνει τέτοιες καταστάσεις. Να σας πω κάτι για την Γερμανία όταν έχουμε 10 cent πτώση στην τιμή του γάλακτος όπως είχαμε ε, στην τελευταία κρίση μιλάμε ανά έτος 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ χαμένα για τους παραγωγούς. Καμία κυβέρνηση του κόσμου δεν μπορεί να μας τα αντισταθμίσει. Είναι λεφτά που λείπουν από τα αγροκτήματα, λείπουν από την ύπεθρα γιατί δεν τα κάνουν μασούροι οι αγρότες, ε, τα δίνουν μετά στην ε, οικονομία. Οπότε αυτό το ένιωσαν όλοι μετά στην αλυσίδα και οι συναλλασσόμενοι με τους αγρότες και όλο. Οπότε η σωστή τιμή και το να προλαμβάνουμε την κρίση είναι η καταλληλότερη ε, λύση. Κάθε λίτρο γάλα το οποίο πηγαίνει στην ε, αγορά ε, απαιτεί να χρησιμοποιηθούν πόροι που από την άλλη πλευρά μπορούν να εγγραφούν αν θέλετε σε ένα θετικό ισοζύγιο για την φύση αν δεν ε, παραγόταν το γάλα. Έχουμε λοιπόν προτείνει και την ε, επέκταση των αρμοδιοτήτων ε, του παρατηρητηρίου της αγοράς γάλακτος, κάτι το οποίο εγκρίθηκε, αλλά όχι σε όλους τους τομείς. Απευθύνω λοιπόν έκκληση στους συναδέλφους στην Επιτροπή Γεωργίας, ειδικώ ε, στις διαπραγματεύσεις για το στρατηγικό σχέδιο, να μην το χάσουμε στόχο, γιατί τώρα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μια καλή λύση για ολόκληρο τον ε, κλάδο και συμφέρουσα. Και μετά μιλάμε συνεχώς για κρίσεις. Εντάξει, διακυμάνσεις υπάρχουν, αλλά τόσο μεγάλες κρίσεις που πλέον δεν αφήνουν τη δυνατότητα να βγάλει τα λεφτά του ο αγρότης ε, δεν είναι δυνατόν και ε, τέλος μια ερώτηση πότε θα κάνετε την εκδήλωση μαζί με τους Αφρικανούς συναδέλφους σας σας ευχαριστώ ο κύριος ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω πως η κυρία Σράιερ, Μαγκίνες και οι υπόλοιποι εδώ πέρα είναι από τους πιο ενεργούς στην Επιτροπή αλλά και η πράσινη ομάδα βεβαίως ενδιαφέρεται και εκπροσωπείται. Σας ευχαριστώ για αυτά τα οποία είπατε. Εγώ είμαι πρώτα αγρότης και μετά βουλευτής. Εκπροσωπώ λοιπόν πολίτες, αλλά ειδικά τους αγρότες. Είμαι σκιώδης συγητής επίσης για την κοινή οργάνωση της αγοράς και μπορώ να σας πω πως μέρη των προτάσεών σας ε, είναι ήδη προς συζήτηση και υπάρχουν οι δυνατότητες να υπάρξει κάποια πλειοψηφία και σας ε, ευχαριστώ για την ε, υποστήριξη. Το βασικό πρόβλημα το οποίο μας ε, εμποδίζει είναι η κατεύθυνση της πολιτικής μας η οποία είναι προς την παγκόσμια αγορά. Αυτό το δόγμα δυστυχώς δεν θα μπορέσω να το αλλάξω και εγώ και οι συνάδελφοί μου. Και αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα το που μας εμποδίζει δηλαδή να δούμε γιατί δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε το κόστος παραγωγής και στο μέλλον. Το ερώτημα λοιπόν είναι μήπως θα πρέπει να μειωθεί η συνολική παραγωγή στην Ευρώπη για να περιοριστούμε στην ευρωπαϊκή αγορά ή μήπως στο μέλλον να τρέφονται τα μοσχάρια ε, μεγάλα αντί να πηγαίνουν στην Ισπανία και στην Ιταλία για να τρέφονται με φινικέλαιο το οποίο εισάγουμε από την Ινδονησία και κόβουμε τα δάση. Μήπως λοιπόν τα, τις αγελάδες, εάν θέλουμε πρωτεΐνες, να τους δίνουμε ψυχανθή αντί για σόγια που εισάγουμε από την Βραζιλία, κάτι το οποίο απαιτεί εκατομμύρια εκτάρια γης και ουσιαστικά την επιδοτούμε εμείς ε, και θα πρέπει επίσης ε, να εστιάσουμε στην ποιότητα και τις ε, ιδιαιτερότητες της ευρωπαϊκής γεωργίας. Γιατί έχουμε αγελάδες ελευθέρας βοσκής, γιατί έχουμε ιδιαίτερα ψηλές ποιοτικέ προδιαγραφές, γιατί τα ζώα έχουν κάποια σημασία για τους Ευρωπαίους πολίτες, γιατί βασιζόμαστε στο ε, Σανό και στο να βοσκάνε οι αγελάδες, κάτι το οποίο επίσης είναι μια αποτελεσματική μέθοδος δέσμευσης ε, του διοξιδίου του άνθρακα. Θα πρέπει λοιπόν για όλα αυτά τα οποία παρέχουν στην κοινωνία οι αγρότες ε, να πληρώνονται κιόλα. Σας ευχαριστούμε κύριε Βάιτς. Εμείς στην Ισπανία δεν ε, ε κτρέφουμε με φινικέλαιο τα ζώα μας και έχουμε αυτή την τύχη. Αλλά, και θα ήθελα να διεκδικήσω εδώ το, τη μεγάλη και πολύ καλή προσπάθεια που κάνει οι τρόφι. Ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τους φιλοξενούμενους. Ήθελα να πω ότι δεν έχετε σωστές πληροφορίες να αφορά τη τιμή του γάλακτος. Η τιμή στη Ρουμανία όπου πωλείται το γάλα 0,23 σεντ. Μπορούμε να καταλάβουμε τα προβλήματα. Καταλάβετε τι προβλήματα έχουμε στο ευρωπαϊκό, ε, ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξέρω, ότι δεν συμμετέχει στην οργάνωσή σας η Ρουμανία, οπότε δεν ξέρετε τα δικά μας στοιχεία, τα στοιχεία για τη χώρα μας. Ο τομέας του γάλακτος πολύ συχνά συζητήθηκε σε αυτή την Επιτροπή Γεωργίας και ανησυχώ πολύ για τη μοίρα του τομέα. Είναι σημαντικός ο ρόλος σας όσον αφορά την επίλυση των προβλημάτων. Όμως ταυτόχρονα είσαστε υπεύθυνοι και για αυτό που συμβαίνει στον τομέα των γαλακτοκομικών. Γιατί το λέω αυτό. Και θα αναφέρω κάτι που αναφέρθηκε και πριν. Η, η, που δίδεται για να μην παράγουν οι γεωργοί. Γιατί να μην οδηγηθούν προς ένα μείγμα ε, παραγωγής, να κινηθούν και προς την παραγωγή κρέατος ταυτόχρονα, διότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, μπορεί να περάσει κανείς από το γάλα στο κρέας. Σίγουρα υπάρχουν πολλά είδη αγελάδων. Μπορεί κανείς να περάσει προς την κτηνοτροφία με ζώα, ε, ανατρέφοντας ζώα για παραγωγή ε, κρέατος. Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Με τα ίδια χρήματα που δίνετε για να μην παράγετε το γάλα, μπορείτε να δώσετε τα χρήματα για την παραγωγή κρέατος. Μετά ήθελα να ρωτήσω, γιατί να μην τονώσετε την μεταποίηση του γάλακτος στις ίδιες εκμεταλλεύσεις. Εχθές πήγα σε εκμεταλλεύσεις επιχειρήσεις του τομέα βοήου και ε, υπάρχει δυνατότητα μεταποίησης και μπορούν να πολλούν τα προϊόντα τους οι γεωργοί πολύ κοντά να, να γίνεται μεταποίηση, να παράγονται φρέσκα προϊόντα και σε τιμές που τους επιτρέπουν να επιβιώσουν. Γιατί δεν προωθείται αυτή η προσέγγιση και όσον αφορά το τομέα του ε, βοηού γάλακτος. Τώρα για τα παραποιημένα προϊόντα. Έχουμε ένα πρόβλημα, τουλάχιστον στην Ανατολική Ευρώπη, που συνδέεται με προϊόντα ε, τα οποία είναι παραποιημένα. Ε, για τυρί, που δεν παράγεται από γάλα φερρυπίν, αλλά με φινικέλαιο. Ε, και αυτό θα πρέπει να εξεταστεί. Να υπάρχουν ειδικέ δομέ στα κράτη-μέλη για να μειωθεί αυτό το φαινόμενο. Αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να επιληθεί, να, μη, να μην επιληθεί, να μειωθεί. Μόνο μαζί μπορούμε να κινηθούμε για να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα μην ρίχνετε τις ευθύνες στο Κοινοβούλιο. Εμείς μόνοι μας δεν μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα, αλλά μπορούμε να το κάνουμε όλοι μαζί, μαζί σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φλάνναγκαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ήμουνα εκτός της θύρας όταν έμπαινα και από, και από τα βασικά γερμανικά που καταλαβαίνω και, και όλα αυτά που λέγατε μόνο αυτά καταλάβαινα. Κύριε Φλάναγκα, πλησιάστε λίγο στο μικρόφωνο γιατί δεν σας ακούνε οι διερμηνείς. συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την παρουσίασή σας. Ερχόμουν, έμπαινα στην πόρτα όταν κάνετε τα σχόλιά σας για την έλλειψη ευρωβουλευτών. Έλλειψη παρουσίας ευρωβουλευτών και νομίζω ότι οι επικρίσεις σας είναι άκρως δικαιολογημένε και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι οι ευρωβουλευτές που είναι εδώ είναι εδώ και μπορούν να είναι εδώ μόνο ε, μία φορά και βλέποντας εδώ βλέπω ευρωβουλευτές που είναι σχεδόν πάντα παρόντες. Αλλά νομίζω ότι οι επικρίσεις σας είναι απόλυτα, απόλυτα δικαιολογημένες. Το είπα αυτό επανειλημμένα σε αυτή την Επιτροπή και χαίρομαι όλος ιδιαίτερος που κάποιος μπαίνει εδώ και τα λέει ομά και σταράτα. Πρέπει να μας το υπενθυμίζετε αυτό. Κάποιοι λένε ότι υπάρχουν άλλες επιτροπές, άλλες συνεδριάσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα. Πώ θα μπορούσε να είναι κάτι πιο σημαντικό από αυτό το γεγονό. Είμαι πλήρε μέλο τη Επιτροπή. Και όταν λειτουργεί και συνεδριάζεται πρέπει να είμαι εδώ. Και αν κάποιο προσβάλλεται, λοιπόν πηγαίνετε, μιλήσετε με του ευρωβουλευτέ που, που σπανιότατα έρχονται εδώ και οι οποίοι δεν είναι ποτέ εδώ. Διότι πληρώνονται πολύ καλά για να το κάνουν. Και σίγουρα περνάνε καλύτερα από τους γαλακτοπαραγωγούς και σίγουρα δεν πάνε το βράδυ στο σπίτι τους με πονεμένες πλάτες από τον κάματο της ημέρας. Άριστα, πολύ καλά κάνατε και τα είπατε αυτά που είπατε. Είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που άκουσα ποτέ σε αυτή την επιτροπή, γιατί αληθεύει. Η παρουσίασή σας ήταν άκρως ενδιαφέρουσα, έχω κάποιες απόψεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει η παραγωγή ε, σωστή, να μην υπάρχει υπερβολικό φωτισμό τη αγορά και θα πρέπει το παρατηρητήριο να δεύτερη φάση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγχει την αγορά και αυτό ίσω να είναι αναγκαίο. Αλλά σε αυτή τη φάση ο γαλακτοπαραγωγό έχει ήδη υποστεί το κόστο τη παραγωγή. Επίση πιστεύω ότι οι γεωργοί θα πρέπει να απαιτήσουν οι συμβουλευτικέ υπηρεσίε να λειτουργήσουν για αυτού και όχι για τι παγκόσμιε πολυεθνικέ. Διότι κάθε αύξηση στην παραγωγή μόνο του μεταπητέ βολεύει. Θα πρέπει να σκεφτούν μόνοι του τι πρέπει να κάνουν οι γεωργοί Μία ερώτηση. Πιστεύετε ότι οι τομέα μεταπίσεω αγροτικών προϊόντων και οι συμβουλευτικέ υπηρεσίε εξυπηρέτησαν του γεωργού και του οδήγησαν μήπω σε ανεξέλεγκτη ε, αύξηση, μήπω θα πρέπει να πιάνουν ανεξάρτητη παραγωγή και να παράγουν για κέρδο. Ε, τι σκέφτεστε για εταιρείε που αγοράζουν γάλα από του γαλακτοπαραγωγού και διατείνονται ότι κατά κάποιο τρόπο βοηθούν την αγροτική κοινότητα αλλά μετά διοχετεύουν, ρουφάνε τα, τα κέρδη τους και τα περνάνε μέσω Λουξεμβούργου για να μην πληρώσουν φόρο, όπως το κάνει μετά στην Ιρλανδία. Και αυτά τα χρήματα τελικά δεν καταλήγουν στη χώρα μας και καταλήγουν τα χρήματα στα χέρια, να το πούμε ειλικρινά, των γκάγκστερ, των συμμοριών. Ποια είναι η άποψή σα για αυτή τη μεθοδολογία όσον αφορά τον τρόπο αντιμετωπίσεω των γεωργών τη εταιρεία. Τελευταία ερώτηση. Είπατε ότι υπάρχουν εκατοντάδε τόνοι γάλακτο σε σκόνη σε παρέμβαση. Ε, και θα ήθελα μια επεξήγηση από αυτά που είπε ο Φιλ Χόγκαν. Είχα καταλάβει ότι το γάλα σε σκόνη είχε πολιθεί. Μπορεί κάποιο να το ξεκαθαρίσει αυτό και να μα εξηγήσει επακριβώ ε, ποια είναι η κατάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συνεχίστε να λέτε αυτά που λέτε. Δεν χρειάζεται να ζητήσετε συγγνώμη από εμά για τίποτα. Καλά τα κάνετε. Ευχαριστούμε κύριε Φλάναγκα. Κύριε Ριβέρα έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τους καλεσμένους μας και να ζητήσω συγγνώμη που καθυστέρησα λίγο. Αλλά είχα συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Γι' αυτό απουσίαζα στην αρχή της συνεδρίασης. Πάντως, έχουμε ήδη σε προηγούμενες συνεδριάσεις αναλύσει τα έγγραφά σας και τις προτάσεις του προγράμματός σας. Με ενδιαφέρει αυτό το ζήτημα της ρύθμισης της αγοράς γάλακτος και των τιμών γάλακτος. Και γι' αυτό είναι πολύ ευπρόσδεκτες οι προτάσεις σας. Έχουμε πάντως κάποιες επιφυλάξεις και αμφιβολίες που θα ήθελα να διασκεδάσετε. Εσείς, πώς συνδέεται αυτό τον οργανισμό παρακολούθησης με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Γάλακτος. Ε, πώς κρίνεται τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητήριου Γάλακτος σε ό,τι αφορά την πρότασή σας που στηρίζεται στο δίκτυο 100, δηλαδή ε, στη σχετική ισορροπία της εθνικής αγοράς, από ό,τι κατάλαβα τουλάχιστον. Πώς λοιπόν θα ορίσουμε αυτό το δίκτυο εθνικής αγοράς και υπό ποιες ε, περιστάσεις. Γιατί στη Πορτογαλία και κατά στην ακόμη χειρότερη Αζόρες η ε, τιμή γάλακτος που πληρώνουμε στον παραγωγό είναι η τιμή κρίσης. Η παραγωγή λαμβάνουν ε, για το γάλα τους ε, τιμή πολύ χαμηλότερη από τον κοινοτικό μεσόρο. Οπότε πώς θα γίνει ο υπολογισμός του δίκτυ, γιατί αν η περίοδος αναφοράς είναι η σημερινή, τότε θα πληγούν οι αζόρες και η μαδέρα. Θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία στις τιμές. Πώς θα την εξασφαλίσουμε όμως με τον υπολογισμό του δίκτυ για να μην πλήξουμε ακόμη περισσότερο κάποιους γαλακτοπαραγωγούς. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μαγκίνες έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ τους ε, εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Γάλακτος. Το πιο σημαντικό είναι ότι η αντίδραση αγοράς ε, στον έλεγχο της ποσότητας λειτουργεί. Υπάρχει μία ε, θετική επίπτωση που είναι αύξηση των τιμών. Είπατε όμω ότι κάτι τέτοιο προποθέτει μια γραφειοκρατική δομή σε έναν τομέα που απελευθερώθηκε από τι γαλακτοκομικέ ποσοστώσει παρόλο που έχουμε ακόμη κάποιες αρνητικές επιπτώσεις αυτής της κατάργησης των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων. Δεύτερο μου σχόλιο αφορά τους νέους, τους νεαρούς αγρότες. Οι νέοι όταν έχουν επιλογή μπορούν να προβούν σε επιλογή, αν έχουν ένα φάσμα επιλογών. Αν όμως ε, ε, ε, αφήσουμε στη απολυθωμένη την ε, γαλακτοπαραγωγή, τότε δεν θα προσελκύει νέους. Πώς λοιπόν θα περιορίσετε αυτό το φυσικό αίσθητο συντήρησης. Επίσης, η ε, οικονομική θεωρία λέει ότι όταν οι τιμές γάλακτος είναι χαμηλές, ο γαλακτοπαραγωγός αισθηκτοδός θέλει να αυξήσει την ποσόστοση, την παραγωγή του μάλλον, την ποσότητα για να αυξήσει το εισόδημα. Οπότε θα πρέπει να έχουμε κάποια θεμελιώδη στοιχεία αγροτική οικονομία κατά νου μιλούμε για ρύθμιση αγορών. Στην Ιρλανδία ευτυχώ έχουμε λιβάδια, οπότε έχουμε αύξηση τη παραγωγή, έχουμε μια συνεταιριστική δομή του γαλακτοπαραγωγικού τομέα με στενού δεσμού των παραγωγών που είναι μέτοχοι αυτού του συνεταιρισμού, κάτι που δεν ισχύει σε άλλα Έχουν διαφορετική δομή, οπότε θα πρέπει να δούμε και τι διάφορε δομές κόστους. Ε, η δομή τη παραγωγής στην Ιρλανδία είναι διαφορετική από τις άλλες χώρες και ίσως χαμηλότερο το κόστος παραγωγής. Επίσης, πολύ σωστά ο κύριος ε, Νίκολσον είπε ότι η επέκταση του γαλακτοκομικού κλάδου επηρεάζει την κρεατοπαραγωγή. Και επίσης έχουμε παραγωγή και μοσχαριών, όχι μόνο γάλακτος. Και εκεί έχουμε κάποιες προκλήσεις ε, για τη διαχείριση της παραγωγής και αυτές οι προκλήσεις αντιμετωπίζουμε τώρα στην Ιρλανδία. Εγώ βλέπω έτσι τον γαλακτοκομικό τομέα υπό τη σκοπιά και των περιβαλλοντικών θεμάτων που θα είναι οι νέες ποσοστώσεις. Είτε μιλάμε για λιπάσματα, για, για ποιότητα του αέρα. Όλα αυτά θα περιορίσουν την επέκταση της παραγωγής τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Και αυτό το μήνυμα θα πρέπει να το διαβιβάσουμε. Επίσης, χρειαζόμαστε κάποια μέτρα αγοράς όταν πραγματικά υπάρχει μια κρίση που ρίχνει τις τιμές. Και Ίσως ήρθε κάπως αργά το πρόγραμμα, πάντως φαίνεται ότι λειτουργεί και αυτό φάνηκε από την παρουσίαση. Σε ό,τι αφορά το dumping των γαλακτοκομικών προϊόντων, τι ακριβώς εννοείτε, γιατί έχουν καταργηθεί οι εξαγωγικές ε, επιδοτήσεις, οπότε πού βλέπετε εσείς το dumping. Αν υπάρχει αυτή η πρακτική, αν υπήρχε δεν τη γνωρίζω. Σε ό,τι αφορά τα αποθέματα, όντως η Επιτροπή μείωσε αισθητά τις ποσότητες ε, 374.000 ε, ε, τόνοι πουλήθηκαν σε πληστηριασμό και 100 μόνο έμειναν στην αποθεματοποίηση. Κάτι που δίνει το σήμα, το, την ένδειξη ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι τιμές και ήδη έχουν αυξηθεί. Εγώ ως ευρωβουλευτής εκπροσωπώ τους ψηφοφόρους μου. Δεν ε, είμαι απουσιολόγος και δεν σημειώνω ποιος παρακολουθεί και ποιος απουσιάζει από την συνεδρίαση. Ε, σέβομαι τα σχόλιά σας για, το, για την προσέλευση, αλλά σε, στο κάτω-κάτω της γραφής όλοι είμαστε υπόλογοι στους ψηφοφόρους μας και αυτή είναι και η ομορφιά της δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαντεκέντελάρη, ο τελευταίος μας ομιλητής. Συγγνώμη αν κατακρεούργησα στην προφορά το όνομά σας. Δεν είναι πρόβλημα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ, όπως και εγώ είμαι στον τομέα του γάλακτο στην Δυτική Φλάνδρα και θα το ξέρετε κι εσείς ότι η περιφέρειά μου είναι πάρα πολύ σημαντική για το γάλα αλλά ακόμη σημαντικότερη για τον ε, τομέα του χοιρινού κρέατος και βεβαίω όπως ξέρετε, και αυτός το τομέα είναι πάρα πολύ ευαίσθητος. Αυτό για να καταλάβετε ότι δεν είμαστε και χτεσινοί, όπως λέμε στα Ολλανδικά. Λοιπόν, για να έχουμε μια ξεκάθαρη συζήτηση, μιλήσατε για επιδοτήσεις και την πλήρη κατάργησή τους. Ε, εδώ πέρα νομίζω ότι είναι σαφώς διχασμένη η άποψη των ε, αγροτών. Ε, δεν ε, έχω πάει ποτέ σε συνάντηση αγροτών που να συμφωνούν σε αυτό κατά πλειοψηφία. Και βεβαίως αυτό αφορά και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ποια είναι η άποψή σας για την ενότητα ας πούμε των αγροτών σε αυτό το θέμα και πως θα έπρεπε να υπάρχει ένα κοινό μέτωπο στο μέλλον. Δεύτερον, για τα μέτρα της ε, κρίσης, εκεί πέρα ήσασταν νομίζω ε, σαφείς για τα μέτρα διαχείρισης κρίσης που έχει η Κομισιόν. Εσείς από ό,τι θέλω, από ό,τι κατάλαβα θέλετε να δημιουργηθεί κάτι το επιπλέον ή θα είναι το μόνο ε, μέτρο διαχείρισης της ε, κρίσης και να μην υπάρχουν τα άλλα μέτρα. Και τέλος, ε, για αυτό το οποίο είπε η κυρία Μπούτα, η αγορά της αποθεματοποίησης, τι μπορεί να γίνει εδώ πέρα ακριβώς για να μπορέσουμε να προσφέρουμε μια καλύτερη απάντηση στην κρίση. Υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε για να διευκολύνουμε την κατάσταση και Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώσαμε το κατάλογο των αγορήτων μας και θα ξαναδώσω το λόγο, θα δώσω μάλλον τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Σκάνελ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να απαντήσουμε ε, στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Γάλακτος, με το οποίο έχουμε συνενθεί πολλές φορές ε, και εκτιμούμε ιδιαίτερο στη συμβολή. Θέλουμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των γεωργών και των γαλακτοπαραγωγών και σίγουρα αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις, ε, ιδιαίτερα τώρα που συζητούμε στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική και του μηχανισμού στήριξη. Συμφωνούμε απόλυτα με τι απόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Γάλακτο για τη σημασία του γάλακτο παραγωγου τομέα και την ενίσχυση των συστημάτων προστασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σα βεβαιώ, κύριε Νίκολσον, ότι αυτό ισχύει και για του άλλου κτηνοτρόφου, όχι μόνο για του γαλακτοπαραγωγού. Δεν ευνοούμε κάποια κατηγορία ει βάρο άλλων. Πάντως, στο παρελθόν είχαμε κάποια μέτρα στήριξη. Είχαμε το σύστημα προαιρετικής μείωσης των ποσοτήτων γάλακτος. Και σίγουρα είχε αισθητή βελτίωση του συστήματος και της ε, επαναφοράς εμπιστοσύνης. Και μάλιστα πρόσφατα στην έκθεση Γεωργίας της ε, Γαλλίας ο Επίτροπος Χόγκαν έλαβε το παράσημο της Λεγιώνας της Τιμής ε, στη Γεωργία ως ε, έμπρακτη αναγνώριση ε, της επιτυχίας του συστήματος της προαιρετικής μείωσης των ποσοτήτων κατά το τέλος της του Επιτροπού Χόγκαν. Επίσης είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι ήταν ένα μέτρο που δεν ε, με σχέση με τις... Ήταν ένα έκτακτο μέτρο σε σχέση με τις δικές σας προτάσεις που έχουν πιο συστηματικά μέτρα. Και αυτή είναι η βασική διαφορά. Το δικό μας ήταν προσωρινό έκτακτο μέτρο ε, και η μετατροπή του σε μόνιμο, κατά τη γνώμη μας, εγείρει πολλά προβλήματα και κινδύνους. Επίσης, ε, ο ρόλος ε, των, ε, της παρέμβασης για την αγορά από βουτυρωμένο γάλακτος σε σκόνη. Τώρα έχουμε 1.300 τόνους, όπως είπε η κυρία Μαγκίνες, το 1 τρίτο δηλαδή, το 1% των αποθεμάτων που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε σίγουρα διαθέσαμε τα αποθέματα, έχουν μείνει ελάχιστα και κατά την αγορά, κατά την ε, θέσπιση της ε, αγοράς είχαμε πολλές επικρίσεις ότι θα καταπιέσουμε τις αγορές, ε, θα, θα μειωθούν οι τιμές, θα είναι αδύνατο να διατεθούν μετά τα αποθέματα. Τελικά ήταν ανεδαφική αυτή η φόβη. Είχαμε αύξηση των αγορών με υψηλότερες τιμές από τις αναμενόμενες με μηδενικό κόστος για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο και μάλιστα αποδείχθηκε ότι αυτό το μέτρο ήταν ε, πολύ επιτυχές για τη σταθεροποίηση των αγορών. Αυτή η παρέμβαση με την αγορά. Επίσης, ό,τι αφορά το dumping των γαλακτοκομικών προϊόντων ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες, απόρριψη μάλλον αυτών των προϊόντων και μαζική εξαγωγή προς, τις, ε, προς την Αφρική και μία αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό το διαψεύδουμε. Δεν έχουμε πια εξαγωγικέ επιστροφέ. Είναι ελάχιστε οι εξαγωγέ μα προ χώρε αυτέ. Οπότε δεν ισχύει αυτό το dumping που είπατε. Παρόλο που εξακολουθεί να μα στοιχιώνει αυτή η κατηγορία ε, και επηρεάζει και την εικόνα και την υπόλοιψη του γαλακτοκομικού κλάδου, ε, εξαγωγής εξαγωγή μα. Παρόλο που είναι πολύ επιτυχημένε οι εξαγωγέ γάλακτο και οι προσπάθειέ μα να αυξήσουμε τι εξαγωγέ δεν ε, ε, υποβοηθούνται αν πρέπει συνεχώ να διαψεύδουμε τέτοιε κατηγορίε ή να πρέπει να τι καταρρύπτουμε. Επαναλαμβάνω, δεν ισχύουν πια, είναι αδεδαφικέ. Και κατηγορηματικά διαψεύδουμε και απορρίπτουμε αυτέ τι κατηγορίε για dumping λόγω εξαγωγικών επιστροφών που δεν ισχύουν πια. Σε ό,τι αφορά την μόνιμη θέσπιση του μηχανισμού σταθεροποίηση, λυπάμαι, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε λίγο πρέπει να αρχίσουμε να περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Περιμένουμε και τον Επίτροπο, τους Επιτρόπους μάλλον. Εντάξει, η Πρόεδρος Μαγκίνες ε, ανακεφαλαίωσε τις αδυναμίες και τους κινδύνους που θα είχε η μονιμοποίηση αυτού του συστήματος παρέμβασης. Εκτός της μεγάλης γραφειοκρατίας που θα ε, αύξανε, θα αυξάνει και το κόστος και σίγουρα από τις άμεσες ενισχύσεις ε, θα έβγαιναν αυτά τα ποσά για τις επιδοτήσεις, άρα οι ίδιοι οι γεωργοί από την τσέπη το πλήρωναν και επίσης ε, θα αμφισβητούνταν έτσι πολύ επιτυχείς μεταρρυθμίσεις ε, που θεσπίστηκαν στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Και για να ολοκληρώσουμε, θα ξαναδώσω το λόγο στα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Γάλακτο. Παρακαλώ όμως τρία λεπτά, όχι παραπάνω. Ο κύριος Ευχαριστώ που μας ε, δίνετε πάλι το λόγο. Θα είμαι σύντομος. Πρώτον, ε, εντάξει, έκανα εγώ μια παρατήρηση στην αρχή, ε, τελείως συναισθηματικά για την απουσία των βουλευτών. Και νομίζω ότι ως πολίτες έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε αυτές τις παρατηρήσεις χωρίς να προσβάλλουμε κάποιον. Δεν ήθελα να προσβάλλω κάποιον. Αλλά όταν μπαίνω και βλέπω αυτά τα πράγματα πρέπει να το πω έτσι λειτουργώ εγώ λοιπόν για τις ε, επιδοτήσεις ε, τα πριν αν έχουμε μια τιμή η οποία καλύπτει το κόστος του γάλακτος δεν χρειαζόμαστε άλλη στήριξη και στόχος πρέπει να είναι αυτά τα 43-45 cent να τα επιτύχουμε και μπορούμε να το επιτύχουμε αν ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα και τότε δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και εάν το εξηγήσετε αυτό στους αγρότες σας, στην Ιρλανδία, στην Ολλανδία, οπουδήποτε, για να φτάσουμε την τιμή του κόστους ε, και τότε δεν θα υπάρχει άλλη επιδότηση νομίζω δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα γιατί και ο καταναλωτής ε, μας βλέπει ως ανθρώπους οι οποίοι λαμβάνουμε επιδοτήσεις δεν το θέλω, δεν το θέλουν και οι ε, συνάδελφοί μου θέλουμε μια λογική τιμή γι' αυτό έχουμε αυτά τα μέτρα Γι' αυτό ξαναλέω πρέπει από κοινού να βρεθεί ένας τρόπος πώς θα ξεφύγουμε από αυτό το δίλημα. Και ακριβώς θα έρθουμε σε επαφή και με όλους τους ευρωβουλευτές, αλλά κάποια στιγμή πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε ότι έτσι όπως λειτουργούμε αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Αν έρθει αύριο μια άλλη καταστροφή, ένα νέο σκάνδαλο, πρέπει να ξεκινήσουμε ξανά από το μηδέν. Για εμένα η πολιτική πρέπει να δημιουργεί το πλαίσιο για να μην ξαναβρεθούμε σε μια τέτοια κρίση και να έχουμε οικονομική καταστροφή. Αυτό θέλουμε εμεί από τους ε, πολιτικούς υπεύθυνου. Εμείς είμαστε αγρότες η δουλειά με εμένα δεν είναι να κάνω πολιτική. Εγώ αρμέγω γελάδε. ο Μπόρις, ο Ιωάννη ε, από τη Δανία, οι συνάδελφοι. Η δουλειά μας είναι να αρμέγουμε. Αλλά θέλουμε έτσι τις ε, οικογενειακές μας επιχειρήσεις που τι έχουμε εδώ και γενιές και φτιάχτηκαν εδώ και γενιές, μην τα ξαναλέω, θέλουμε να μπορέσουμε να τι παραδώσουμε στα παιδιά μα, να γίνουν μεγαλύτερε. Όχι να είναι καταχρεωμένες. Εάν δεν έχουμε πλέον κάλυψη του κόστους, εμείς οι τέσσερις σε δέκα χρόνια δεν θα ασχολούμαστε, δεν θα υπάρχει κανείς. Θα έρθει εδώ μέσα η Κανόνε, η Καμπίνα, η Νεστλέ και με αυτούς θα μιλάτε. Και θα σας πούνε ποια πολιτική θα πρέπει να κάνετε. Ακόμα υπάρχουν αγρότες εδώ μέσα, αλλά προσεχώς θα υπάρχουν μόνο εκπρόσωποι εταιριών. Σας ευχαριστούμε κύριε Σιώπιος. Σας ευχαριστούμε θερμά και σας συγχαίρουμε για τις προτάσεις σας. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η συζήτηση που είχαμε, όπως είδατε με τη συμμετοχή όλων των παρόντων ευρωβουλευτών. Μία πολύ σύντομη διακοπή ενός λεπτού για να αποχαιρετήσουμε τους καλεσμένους μας και να υποδεχθούμε τους επόμενους μας προσκεκλημένους. Comenzamos. Συνεχίζουμε. Number English too. Comenzamos. Περνάμε στο σημείο 4 της ημέρησης διάταξης προβλέπει την παρουσίαση της τελικής έκθεσης της Ειδικής Ομάδας Εργασίας για την Αγροτική Αφρική. Η παρουσίαση θα γίνει από τον επικεφαλής της ομάδας αυτής, τον κύριο Τόμ Άρνολτ, τον οποίο και καλωσορίζω. Παρουσία του Επιτρόπου Γεωργίας Φιλ Χόγκαν. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Για μια ακόμη φορά στην Επιτροπή Γεωργίας και παρουσία της κυρίας Χωσέφα Σάκο. Καλώς ήρθατε κυρία Σάκο που είναι Επίτροπος Αγροτικής ε, Οικονομίας και Γεωργίας της Επιτροπής Αφρικανικής Ένωσης. Θα δώσω πρώτο το λόγο στον πρόεδρο της Task Force, της ειδική αυτής ομάδας εργασίας για την Αγροτική Αφρική, τον κύριο Τόμ Άρνολτ, που θα μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα αυτής της σημαντικής ομάδας εργασίας. Όπως ξέρετε, ο κύριος Άρνολτ ε, είναι απόφυτος ε, αγροτικής οικονομίας στο University College του Δουβλίνου και έχει μεταπτυχιακό στο Trinity College του Δουβλίνου και στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβάν και επίσης ε, έχει επίτιμα διδακτορικά στα πανεπιστήμια αυτά και στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας. υπηρέτησε σε πολλές κυβερνητικές και μη κυβερνητικές θέσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο είναι ένας ε, αναγνωρισμένου φήμης εμπειρογνώμων και έχει πλούσια πείρα από πολλούς τομείς στις διάφορες αυτές τις θέσεις που υπηρέτησε. Γι' αυτό νιώθουμε ιδιαίτερη τιμή που τον ε, υποδεχόμαστε εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας. Έχετε 10 λεπτά κύριε Άρνολτ για να μας κάνετε την παρουσίασή σας. Κατόπιν ε, τη συζητήσεως θα δευτερολογήσετε για να απαντήσετε στις απορίες. Έχετε 10 λεπτά, καλώς ήρθατε και πάλι και σας ακούμε. thank you. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το θερμό καλωσόρισμα που συνεχίζει τις επαφές μας μετά τον Νοέμβριο που επίσης ε, είχα τη χαρά να λάβω το λόγο στην Επιτροπή. Τότε βρισκόμαστε στα μέσα της δουλειάς της Task Force. Τώρα με μεγάλη χαρά και τιμή θα σας παρουσιάσω την τελική έκθεση αυτής της ειδικής ομάδας εργασίας που εμ, επίσημα παρουσιάστηκε πριν από μία μόλις ώρα από τον Επίτροπο Χόγκαν και την Επίτροπο Σάκο. Πριν περάσω στο περιεχόμενο της έκθεσης, θα ήθελα να κρατήσετε όλοι έναν αριθμό. 800 εκατομμύρια. Αυτός είναι ο αριθμός των ανθρώπων που θα μπουν στην αγορά εργασίας της Αφρικής τα επόμενα 30 χρόνια. Και είναι οι άνθρωποι που θα είναι μεταξύ 15 και 64 ετών τα επόμενα 30 χρόνια. Μεταξύ του 2020 και του 2050 η Αφρική ε, θα αντιπροσωπεύει τα τρία τέταρτα της αύξησης της παγκόσμιας, του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού. Και αυτή η αύξηση του εργατικού δυναμικού συνδέεται φυσικά με την αύξηση του πληθυσμού. Ο πληθυσμός της Αφρικής διπλασιάστηκε τα τελευταία 30 χρόνια και πρόκειται να ξαναδιαπλασιαστεί την επόμενη τριακονταετία. Μέχρι το 2050 η Αφρική θα αριθμεί περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πώς λοιπόν θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και εισόδημα ώστε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες αυτού του αυξανόμενου εργατικού δυναμικού και του αυξανόμενου πληθυσμού. Αυτό είναι από τις σημαντικότερες ε, πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις των καιρών μας. Και για να ε, ανταπεξέλθουμε σε αυτή την πρόκληση θα πρέπει να μετασχηματιστεί τελείως η αφρικανική οικονομία και να αξιοποιηθεί στο έπακρο ο αγροδιατροφικός κλάδος και η αγροτική οικονομία. Και γι' αυτό στην έκθεση προτείνουμε διάφορες ιδέες και συστάσεις που πιστεύουμε ότι θα οδηγήσουν στην αξιοποίηση αυτού του μεγάλου δυναμικού της Αφρικής για μεταμόρφωση. Επίσης εξετάζουμε την μεγάλη ποικιλομορφία της Αφρικής ό,τι αφορά την οικονομική της ανάπτυξη και ζητούμε μαζικές ε, και μακροπρόθεσμες επενδύσεις ε, στην ε, διατροφή, στην παιδεία, στην υγεία των Αφρικανών και στην περιορισμό των διενέξεων στην Αφρική, κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και επιτακτική ανάγκη αν θέλουμε πραγματικά ανάπτυξη στην Ήπειρο αυτή. Και όταν επανερχόμαστε στο βασικό μας στόχο, στον αγροδιατροφικό κλάδο και την αγροτική οικονομία, εκεί κάνουμε κάποιες συστάσεις σε ό,τι αφορά τη στρατηγική και τις πολιτικές που θα πρέπει να εφαρμοστούν. Και επίσης λέμε πώς θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Ε, διαδικασία και εταιρική σχέση που χρειάζονται για την υλοποίηση αυτού του μετασχηματισμού στην Αφρική. Σε ό,τι αφορά τις ανάγκες, προτείναμε έξι βραχυπρόθεσμες πρωτοβουλίες προκειμένου να ε, διασφαλιστούν θετικά αποτελέσματα και τέσσερις στρατηγικούς κλάδους δράσης που εφαρμόζονται πιο μέσο και μακροπρόθεσμα. Το πακέτο των βραχυπρόθεσμων μέτρων περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενό καινοτόμου προγράμματο τοπική δράση που θα προσαρμόζεται στι αφρικανικέ περιστάσει, fast track για τη χρηματοδότηση των σχεδίων που αφορούν τη διατροφή και τα σχεδίων κλιματική δράση, επέκταση της στήριξη το, ε, περιφερειακού εμπορίου και της ε, ολοκλήρωσής του και τα συστήματα ασφάλειας των τροφίμων καθώς και αδελφοποίησης και προγράμματα ανταλλαγών. Σε ό,τι αφορά του ε, τέσσερι στρατηγικού τομεί που αναπτύσσονται στα αριθμα κεφάλαια, καταρχήν μια περιφερειακή προσέγγιση στο σχεδιασμό το, της δημιουργίας θέσεων και αύξηση του εισοδήματο την ανάγκη ε, δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε ό,τι αφορά την παροχή βασικών υπηρεσιών σε μικρομεσαίες πόλεις και στην Ήπεθρο. Επίσης, ε, υπό το φως της αγροτικής ανάπτυξη θα πρέπει να ληφθούν όλα αυτά βιώσιμη διαχείριση το, της γης και των ε, φυσικών πόρων, καθώς και των κλιματικών δράσεων. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την κλιματική δράση για να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα απέναντι στις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών. Ε, μάλιστα, η Αφρική είναι ιδιαίτερα ευάλωτη και θα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στο μέλλον στι κλιματικέ αλλαγέ. Τρίτον, βιώσιμο μετασχηματισμό τη Αφρικανική Γεωργία. Προτείνουμε μέτρα για την υλοποίηση άμεσης ανάπτυξης, γεωργικής ανάπτυξης, χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερο στόχο της, την οικογενειακή εκμετάλλευση, την οικογενειακή γεωργία, δημιουργώντα ε, ικανότητε ε, ε, στι οργανώσει παραγωγών και επίση θα πρέπει να αναπτύξουμε τι τοπικές αγορές παραγωγή τροφίμων και το κλάδο, αυξάνοντα επενδύσεις. Ε, τις προδιαγραφές ασφάλειας και ενισχύοντας το ενδοαφρικανικό εμπόριο στα γεωρικά αγαθά και τρόφιμα. Αυτό είναι σημαντικό δυναμικό που θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Θεωρούμε ότι τέτοιε βραχυπρόθεσμε και μακροπρόθεσμε πράξει ε, είναι απαραίτητε για τη μεταμόρφωση, αλλά θα μπορούσε και η Ευρώπη να συμβάλλει με την εμπειρία τη ε, από τα όσα έχουν συμβεί στην Ευρώπη, αλλά και στα πλαίσια τη ευρωαφρικανική συνεργασία που έχει ήδη Πολύ χρόνια εφαρμογή. Και τώρα περνάω στο πώ θα υλοποιήσουμε αυτό το μετασχηματισμό. Η βασική μα σύσταση για το πώ θα πρέπει να υλοποιηθεί αυτό ο μετασχηματισμό είναι η εφαρμογή καινοτόμα εταιρική σχέση για μια ανάπτυξη χωρί αποκλεισμού του αγροδιατροφικού κλάδου τη Αφρική και τη αγροτική οικονομία. Μια τέτοια εταιρική σχέση θα εδράζεται σε αφρικανική πολιτική ηγετική θέση που θα υποβοηθάτε από την ε, εμπειρογνωσία, την πείρα και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να έχει ηγετική θέση πολιτική Αφρική με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρία επίπεδα. Διαπροσωπικό, διεπιχειρησιακό και διακυβερνητικό και επίσης ε, μακροπρόθεσμο χαρακτήρα με, με διάλογο πολιτικής, ε, με πολιτική συνέπεια και από τις δύο πλευρές και την υποστήριξη των θεσμών που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή χρηστών πολιτικών. Και έρχομαι στα συμπεράσματα τώρα. Ε, προσπάθησα ε, σε αυτή τη σύντομη παρουσίαση να συνοψίσω την πολυσέλιδη έκθεσή μου και να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Τρεις είναι οι βασικές ιδέες. Καταρχήν, θα πρέπει να έχουμε μια διαπαιδαγωγική διαδικασία. Μην ξεχνάτε ότι 800 εκατομμύρια άνθρωποι θα ε, εμπλουτίσουν το, το εργατικό δυναμικό της Αφρικής τα επόμενα 30 χρόνια. Θα πρέπει αυτό το σημαντικό στατιστικό στοιχείο να ληφθεί υπόψη και να εδρεωθεί στην πολιτική και δημόσια σκέψη στην Ευρώπη και στην Αφρική. Και επίσης θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την επιτακτική ανάγκη της εξασφάλιση, βράχη και μακροπρόθεσμων πολιτικών για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της αύξησης και της εργασίας και του εισοδήματος για τέτοιο αυξανόμενο εργατικό δυναμικό και αφρικανικό πληθυσμό. Επίσης, η έκθεση αυτή δημοσιεύεται ε, μια εποχή που φαίνεται ότι υπάρχει πολιτική βούληση υλοποίησης αυτών των συστάσεων η Επίτροπος Σάκο και η Επίτροπος Χόγκαν μας υποστήριξαν στο έργο μας. Οπότε το θεμελιώδες ερώτημα είναι τώρα. Μπορεί αυτός ο προφανής ενθουσιασμός των δύο επιτρόπων και η δέσμευσή τους να συνοδευτεί από τον αντίστοιχο ενθουσιασμό των Υπουργών Γεωργίας και ακόμη πιο σημαντικά από την δέσμευση των Υπουργών Οικονομίας και των αρχικών κρατών και κυβερνήσεων. Ένα σημαντικό πρώτο βήμα θα μπορούσε να είναι η υλοποίηση των βραχυπρόθεσμων μέτρων που προτείνουμε στην έκθεση, στα πλαίσια ενός σχεδίου δράσης και μιας νέας συμμαχίας ευρωαφρικανικής για βιώσιμες θέσεις απασχόλησης. Και αυτό θα μπορούσε να συμφωνηθεί στην επόμενη ε, συνάντηση των Ευρωαφρικανών Υπουργών Γεωργίας τον Ιούνιο. Τέλος, στην έκθεσή μας ζητούμε ένα αυρο, ευρωαφρικανικό θεματολόγιο για, για τον ακροτικό μετασχηματισμό και προτείνουμε ένα μενού πολιτικής που θα πρέπει να προσαρμόζεται στι τοπικέ εθνικέ και περιφερειακές περιστάσεις. Επίσης, ε, ε, επισημαίνουμε την ανάγκη του να δώσουμε στον αγροδιατροφικό κλάδο και την αγροτική οικονομία κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών και εντό Αφρική και μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρική για να ευοδοθεί αυτή η εταιρική σχέση. Και θα ολοκληρώσουμε την τελευταία ε, γραμμή της εκτελεστικής μας έκθεσης ε, που λέει ότι θα θέλαμε να βάλουμε τη συνεργασία στον ακροδιατροφικό και τον γεωργικό κλάδο στο επίκεντρο, στην καρδιά των σχέσεων μεταξύ των δύο υπήρων μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Αρνόλτ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η κοινή συνεδρίαση που είχαμε οι Επιτροπές Γεωργίας και Ανάπτυξης στις 21 Νοεμβρίου του 2018 ε, Είχατε έρθει και μα ενημερώσετε, κύριε Άρνολτ, για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ειδική ομάδα εργασία. Και τώρα που μας παρουσιάσετε και τα τελικά συμπεράσματα, την τελική έκθεση, διαπιστώσαμε ότι όντω ε, ε, γίνεται μεγάλε προσδοκίε. Θα πρέπει να μην διαψευστούν τώρα και να γίνουν τα απαραίτητα διαβήματα που απαιτούνται όχι μόνο από την Επιτροπή και από τους δύο αλλά και από τις κυβερνήσεις των ε, διαφόρων χωρών και της Ευρώπης και της Αφρικής. Δυστυχώς αυτή τη φορά σήμερα δεν μπορέσαμε να οργανώσουμε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Άγκρη και ΔΕΒΕ, αλλά καλέσαμε τα μέλη της Επιτροπής ΔΕΒΕ στην σημερινή μας συνεδρίαση. Ξέχασα να καλωσορίσω αυτά τα μέλη όταν ε, ξεκινήσαμε τη συζήτηση, θα το κάνω τώρα και να δώσω το λόγο στον αρμόδιο Επίτροπο Γεωργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Φιλ Χόγκαν, για πέντε λεπτά όμως παρακαλώ. Έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ τους κυρίους και κυρίες. Ευχαριστώ που οργανώσατε την εκδήλωση. Χαίρομαι που έχουμε την Επίτροπο της Αφρικής Ενώσεων για Γεωργία, την κυρία Σάκο και τον Τόμ Άρνολτ που είναι υπεύθυνο για Task Force, Task Force, για να σα ενημερώσουμε για τι εργασίε τη ομάδα εμπειρογνωμόνων και που συνέταξε αυτή την έκθεση 71 σελίδων αφορά ανθρώπους, το λαό της Αφρικής, του λαού της Αφρικής και της Ευρώπης, αφορά πολιτικούς επιχειρηματίες, επαγγελματίες του αγροτροφημικού τομέα και κυρίως για τους πολίτες της υπαίθρου που συνεργάζονται για αμοιβαίο συμφέρον σαν ισότιμοι πολίτες. Είναι πολύ σημαντικό το ότι η Επιτροπή ε, Ανάπτυξης και η Γεωργική Επιτροπή συνεδριάζουν μαζί για να μπορέσουν να συνεδριάσουν από κοινού τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικανικής Υπήρου. Και χαίρομαι που μοιράζομαι τη σκηνή με αυτούς που ήταν υπεύθυνοι σε μεγάλο βαθμό τόσο ώστε να δώσει καρπούς η προσπάθεια. Αυτή η ομάδα κρούσης δημιουργήθηκε μια κρίσιμη στιγμή όσον αφορά ε, τη νέα Συμμαχία Αφρική και Ευρωπαϊκή Ένωση για βιώσιμη ανάπτυξη και θέσει εργασία. Είναι η πρώτη έκθεση που δίνει συγκεκριμένε συστάσει πολιτική ε, για αυτό το σκοπό. Με αυτές τις στάσεις τώρα έχουμε δικό χάρτη για τον αγροτροφωμικό τομέα και την Ήπεθρο για τις δύο υπήρους. Όταν δημιουργήσαμε την Task Force ζητήσαμε η ομάδα να γεφυρώσει το κενό μεταξύ ευκαιρία και πραγματικότητα και χαίρομαι που λέω ότι η έκθεση τελικά πέτυχε αυτό που θέλαμε να πετύχει. Πρόθεσή μας δεν είναι να λέμε απλώς λόγια αλλά να δράσουμε και δεν πιστεύω να ετοιμάζουμε μια ομάδα εμπειρογνωμών που συντάσσει μια έκθεση μετά σκονίζεται. Το κάναμε. Αυτή η Task Force έδωσε τελικά ρηξικέλευθες ε, νομοθεσίες όσον αφορά την παραγωγή τροφίμων και ελπίζω ότι τελικά θα μπορέσουμε να κάνουμε και τώρα με αυτή την έκθεση τελικά θα μεταφραστεί σε πρωτοβουλίες και πολιτική με νόημα. Η έκθεση Task Force μας ζητά να περισσότερα, καλύτερα και διαφορετικά ε, και πρόσδεκτο το αίτημά τη για μια δαφική προσέγγιση στην ανάπτυξη τη υπαίθρου. Η δική μα εμπειρία στην Ευρώπη καταδεικνύει ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Επίση, καλωσορίζω το ότι τονίζει τη σύμπραξη μεταξύ Ευρώπη και Αφρική σε τρία επίπεδα, όπω είπε ο Πρόεδρο, λαοί με, λαού, με λαού, επιχειρήσει με επιχειρήσει, κυβερνήσει με κυβερνήσει. Η λογική δράση μεταξύ των κοινωνιών μα, επιχειρήσεων και κυβερνήσεων είναι το κλειδί, ούτω ώστε να έχουμε τελικά αποτελέσματα. Αυτή είναι καλύτερη προσέγγιση από τη συνεργασία που κάνουν άλλε χώρε. Ιδιαίτερα καλωσορίζω τη εστιάζεται έκθεση στο πόσο ο ιδιωτικό τομέα μπορεί να παράσχει υπεύθυνε επενδύσει, ούτω ώστε να πετύχουμε στρατηγικέ για τον αγροτροφημικό τομέα και θέσει εργασία για την Αφρική και να βοηθήσουμε σε θέματα ασφαλεία τροφίμων. Θα θέλω να τονίσω κάποιε συγκεκριμένε δράσει, οι οποίε ε, αναφέρθηκαν. Η πρώτη δράση. Ταμείο και συμφωνήθηκε η χρηματοδότηση για τα αγροτροφομικά και με την Γαλλική Αναπτυξιακή Υπηρεσία θα συνεργαστούμε. 85 εκατομμύρια ευρώ είναι σε ποσά για εγγύησει και 8,5 εκατομμύρια ευρώ σε τεχνική αρρωγή. Ε, το Ταμείο θα βοηθήσει να διευκολυνθεί η δανειοδότηση και να υπάρχει μόχλευση όσον αφορά τι ιδιωτικέ επενδύσει στην Αφρική, όσον αφορά τον αγροτροφημικό τομέα. Αυτό το ταμείο ταιριάζει πολύ καλά με δράσει που ξεκινήσαμε να ενισχύσουμε τι οργανώσει των ε, γεωργών. Το Ταμείο ξεκίνησε πριν από δύο εβδομάδε και διευκολύνει τι οργανώσει ε, των γεωργών και του συνεταιρισμού να έχουν καλύτερη πρόσβαση στο κεφάλαιο. Και αυτό θα είναι υποφελέ για τα μέλη και θα υπάρξει βιώσιμη επένδυση που χρειάζεται και η ε, Αφρικανική Ένωση και θέλει να προωθήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ορίζεται η πρόταση επίση για ένα ε, πρόγραμμα στην Αφρική που δημιουργήσει απασχόληση και θα αναπτύξει την Ήπεθρο. Ε, θα συμμετέχουν οι τοπικοί φορεί και τελικά θα εμπνευστούν από το πρόγραμμα Leader, την κάτωθεν προσέγγιση, όπω το ευρωπαϊκό Leader. Θέλουμε να προωθηθεί γρήγορα. Θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση μεταξύ ευρωπαϊκών ομάδων Leader και Αφρικανικών για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και ανταλλαγή πληροφοριών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να παράσχει υποστήριξη για να δημιουργηθεί δυναμικό σε τοπικό επίπεδο για τοπική δράση. Και τρίτον, ορίζω την πρόταση του Task Force για προγράμματα αδελφοποίηση θα πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή μεταξύ ε, γεωργών Αφρικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι να εμπνευστούν οι νέοι καλλιεργητές και να μάθουν ένας από τον άλλον, να υπάρχει εκπαίδευση, κατάρτιση και προγράμματα για επαγγελματική κατάρτιση αδελφοποίηση ώστε να επαγγελματοποιηθούν αυτοί που εργάζονται στον τομέα αυτό. Η έκθεση σωστά προβλέπει μεγάλο ρόλο για τον ιδιωτικό τομέα όσον αφορά τη αυτοτική μεταμόρφωση τη Αφρική, κυρίω όσον αφορά την ανάπτυξη του αγροτροφημικού τομέα, εστιαζόμενοι επί ενδογενών μικρομεσών επιχειρήσεων. Έχουμε την πλατφόρμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής ε, για τον τομέα αυτό που θα δώσει ευκαιρίες στην ιδιωτική επένδυση για να δημιουργηθεί δικτύωση μεταξύ των εταιριών της Αφρικανικής Ενώσεως και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της οργανώσεις παραγωγών και στην Αφρική και στην ε, Ευρώπη. Άλλο τομέα όπου μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα μαζί πιστεύω είναι να, να προστατεύσουμε τις ε, γραφικές ενδείξεις των προϊόντων το συστήματά μα για, την, για πνευματικά δικαιώματα τη υπαίθρου που λειτουργήσε καλά για την ύπεθρο στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στατηγικές γεωγραφικέ ενδείξει των προϊόντων τους ώστε να βοηθήσει ε, τα μέλη να προσθέσουν ε, αξία στα προϊόντα που παράγουν. Οπότε υποστηρίζουμε πλήρω αυτή την πρωτοβουλία τη Αφρικανική Ένωση και θέλουμε να κινητοποιήσουμε τα πόρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ υποστήριξη ε, αυτού του εφαρμογή αυτή τη στρατηγική για τη γεωγραφική προέλευση. Και αυτό είναι κάτι που θα λειτουργήσει στου επόμενου μήνε. Τέλο, θα ήθελα να απαντήσω στην έκκληση τη Task Force για να υπάρχει πολιτική, μια συνεχτική πολιτική στον τομέα αυτό συζητείται στην Αφρική το θέμα της αγωγών τροφίμων και κάθε φορά των συγκριωμένων αναγκών ε, των παραγωγών, των τοπικών και των πληθυσμών. Δεν είναι απλό θέμα, αλλά εκεί υπάρχουν προβλήματα. θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελεί τμήμα των λύσεων. Γι' αυτό το λόγο και να εξασφαλίσουμε ανοιχτή και ενταξιακή προσέγγιση όσον αφορά συγκεκριμένε δράσει και επόμενα βήματα που προέρχονται από τι τάσει τη Task Force, η Ευρωπαϊκή Επίτροπη θα ξεκινήσει μια ε, διαδικτυακή διαβούλευση με του ενδιαφερόμενου φορεί τη Αφρική για την έκθεση Task Force και για την προσέγγιση που ακολουθεί η ομάδα αυτή κρούση, ε, λαμβάνοντα υπόψη την κατάσταση που υπάρχει όσον αφορά το εμπόριο, τον αγροτροφημικό μεταξύ των δύο πύρων. Τα αποτελέσματα διαβουλεύσεων τελικά θα τροφοδοτήσουν την, την τρίτη διπουργική διάσκεψη στη Ρώμη ε, που ετοιμάζεται για φέτος τον Ιούνιο με τη συμμετοχή των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικανικής Ένωσης για τα θέματα της ε, γεωργίας. Οπότε χαράζει ένας νέος τομέας όσον αφορά ε, μια νέα εποχή για τις σχέσεις Αφρικής-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο πρόεδρος Γιούνκερ την υποστήριξε και ο πρόεδρος Μακρόν υποστήριξε τη σημασία που έχουν οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και Αφρικής σε πρόσφατη ομιλία του στο Παρίσι για τη Γεωργία. Και τα μέλη αυτής της Επιτροπής των δύο επιτροπών υποστηρίζουν ε, την προσπάθεια και το χαιρετίζω αυτό. Και βασιζόμαστε και στην μελλοντική σα υποστήριξη. Επίση, θα παρουσιάσω αυτή την έκθεση στην, στο Συμβούλιο Υπουργών τον Απρίλιο Γεωργία και Αλία και 21 Ιουνίου Επίτροπο Άκο και εγώ θα ξεκινήσουμε την τρίτη συνεδρίαση Ευρωπαϊκή Ενώσεω Αφρική στη διάσκεψη υπουργική στη Ρώμη πριν από τη διετή διπουργική τη ΦΑΟ. Καλή στιγμή λοιπόν να προωθήσουμε το σχέδιο δράση, να εμβαθύνουμε το διάλογο όσον αφορά τη γεωργική πολιτική και θέλω να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία να ευχαριστήσω την κυρία Σάκο και την ομάδα μα για τι προσπάθειε που καταβλήθησαν για συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ και την ομάδα τη. Αύριο είναι η Διεθνή ημέρα γυναικών, Παγκόσμια ημέρα γυναικών και στην Ήπεθρο οι γυναίκε παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά την ασφάλεια τη διατροφή και τη Ήπεθρου. Παρά τα αυτά δεν έχουν αρκετέ δυνάμει και εξουσίε στα χέρια του και δεν μπορούν να κάνουν επιλογή για τη χρήση των γεών, για τι δαπάνε και τη χρήση των εισοδημάτων. Αυτή η έκθεση τον γνωρίζει και έχει πολλέ πολύτιμε προτάσει να κάνει ώστε να ισχύσουμε τα δικαιώματα των γυναικών ε, αγροτών και θα πρέπει να έχουν ισότιμη ε, πρόσβαση στους πόρους και η έμφυλη διάσταση λαμβάνεται υπόψη όλε τι πολιτικέ. Θα ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα στο Ευρωπαϊκό Ένωση 5 εκατομμυρίων βασισμένο στι φορεί τη Ρώμη στον ΟΗΕ που υποστηρίζουν την ενίσχυση των γυναικών. Το πρόγραμμα θα αντιμετωπίσει τι ανισότητε ε, των φύλων και τις ρίζες των ανισοτήτων και την ύπεθρο και θα γίνει μεταμόρφωση τελικά που θα δώσει δύναμη στις γυναίκες, στις νοικοκυριά, στις κοινότητες, στις κοινωνίες τους ωστόσο να προωθήσουν την ευημερία πάντων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δώσατε να παρουσιάσω αυτή την έκθεση και ευχαριστώ εκ νέου ε, για τις προσπάθειες που καταβάλλετε, την αφοσίωση στο θέμα. Σας διαβεβαιώνω ότι και εμείς θέλουμε να μεταφράσουμε τις συστάσεις αυτές σε πραγματικότητα στην ε, σύμπραξη αυτή Ευρωπαϊκής Ενώσης Αφρικής. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα που μας αναγγείλατε για να προωθήσουμε την ισότητα των φύλων. Και επίσης πολύ επίκαιρο γιατί αύριο εορτάζουμε την ημέρα των γυναικών, την 8η Μαρτίου. Σημαντική μέρα για να διεκδικήσουμε την ισότητα των φύλων. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Επίτροπο Σάκο να σας την παρουσιάσω, να παρουσιάσω το βιογραφικό της. Είναι γεωπόνος η κυρία Σάκο, κορυφαία αγρονόμος στην Αφρική. Τον Ιανουάριο του 2017 εξελέγει Επίτροπος Αγροτικής Οικονομίας και Γεωργίας της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης. Προηγουμένως ήταν σύμβολος στα Υπουργεία Γεωργίας και Περιβάλλοντος της πατρίδας της, της Αγκόλα. Επίσης για τρία χρόνια ήταν Γενική Γραμματέας της Διαφρικανικής Ένωσης Καφέ, ακτή του Ελεφαντοστού και επίσης έχει εργαστεί διεθνώς σε πολυάριθμες περιφερειακές και παγκόσμιες οργανώσεις γεωργίας σε τομείς που υποστηρίζονται μεταξύ άλλων από την Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου, την Αφρικανική Ένωση, την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξη ή τη ΦΑΟ. Επίση συμμετείχε ενεργά σε πολλέ περιφερειακές οργανώσεις με στόχο να αντιμετωπιστούν οι προκλήσει που αντιμετωπίζουν κυρίω οι μικροκαλλιεργητέ στην Αφρική. Πολύ ενδιαφέρον το βιογραφικό και εντυπωσιακό τη ε, κυρία Σάκο, που είναι πραγματικά κορυφαία εμπειρογνώμονα. Τη δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ μιλάω ισπανοπορτογαλικά. Η επίσημη βέβαια, η μητρική μου γλώσσα είναι τα πορτογαλικά, αλλά καταλαβαίνω τα ισπανικά. Θα μιλήσω όμως αγγλικά τώρα. Κυρίες ε, και κύριοι βουλευτές, ε, κύριε Επίτροπε, κυρίες ε, και κύριοι, χαίρομαι ιδιαιτέρως που βρίσκομαι σήμερα σε Βρυξέλλες για την παρουσίαση της τελικής έκθεσης για την ομάδα εργασία για την γεωργία της Αφρικής. Σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Μουσάφα Μουχάχ τον πρόεδρο της Αφρικανικής Επιτροπής. Επίσης, να ευχαριστήσω τον Επίτροπο, τον κύριο Χόγκαν, για την πρόσκληση που με επίφθηνε να σας ε, μιλήσω σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κυριότερος εταίρος μας, ε, είναι γύρω στο 35,7% του αφρικανικού εμπορίου, εισαγωγών και εξαγωγών δηλαδή, το 2017. οι σχέσεις μας έχουν ανθίσει και τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τέρος και σύμμαχος της Αφρικανικής Επιτροπής. Έχουμε μια ταχύτατη αστικοποίηση, αλλά παρόλα αυτά η Ήπειρος εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να είναι υπαίθρια ο πληθυσμό που ζει στην Ήπεθρο μειώθηκε ελάχιστα από το 69% το 2000 στο 61% το 2016. Ε, λοιπόν, βλέπετε λοιπόν πως ε, υπάρχει μια, ένας μετασχηματισμός των αγροτικών κοινοτήτων. Στο συνάντηση υψηλού επίπεδου μεταξύ της ε, Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικανικής Ένωσης στις 23 Μαΐου 2018 εδώ στις Βρυξέλλες και οι δύο πλευρές ενίσχυσαν ε, περαιτέρω την ε, συνεργασία τους και τη μελλοντική εταιρική του σχέση και υιοθέτησαν συγκεκριμένα μέτρα για να δουν κάποια πιεστικά παγκόσμια ζητήματα όπως η ασφάλεια και η ειρήνη, η μετανάστευση, η δημιουργία θέσεων εργασία και η γεωργία. Η πρωτοβουλία αυτή ακολούθησε την δέσμευση που έγινε στην πέμπτη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικανικής Ένωσης στο Αμπιτζάν το 2017 δηλαδή την επέκταση της ε, συνεργασίας στην επιστήμη και την ε, τεχνολογία, την αγροβιομηχανία, την ανανεώσιμη ενέργεια, την πράσινη και την γαλάζια οικονομία, την ε, διακυβέρνηση, τις εκλογές, την ειρήνη και την ασφάλεια. Συγκεκριμένα όσον αφορά την οικονομία της υπαίθρου, συμφωνήσαμε πως η Κομισιόν θα έφτιαχνε μια ομάδα φορολογίας ακριβώς για να δώσει την εμπειρία του και πιθανές συστάσεις ε, στην ε, Κομισιόν της Αφρικανικής Ένωσης στα ζητήματα που αφορούν τη Γεωργία συνολικά. Ξεκίνησε λοιπόν η ομάδα εργασίας αυτή τον Μάιο του 2018 και περιλαμβάνει προσωπικό το οποίο έχει την σχετική εμπειρία στα ζητήματα γεωργίας, αναπτυξιακής πολιτικής ή μετανάστευσης και σχετικά θέματα στον τομέα αυτών της Αφρικής και συναντώνται τακτικά από αρχές ε, Δεκεμβρίου 2018 και εστιάζουν σε ζητήματα εφορίας, δημιουργίας εισοδήματος ε, στον ε, τομέα της αγροδιατροφής. Η συστάση της ομάδας εργασίας είναι να εφαρμοστεί μια καινοτόμως εταιρική σχέση για μια βιώσιμη ανάπτυξη και στην Αφρικανική Ήπειρο λαμβάνοντας υπόψη και την διάσταση του φύλου, όπως ανέφερε και ο συνάδελφος. Ότι δηλαδή θα πρέπει ακριβώς να υπάρχει αυτή η γενική προσέγγιση σε οποιοδήποτε αναπτυξιακό πρόγραμμα στην Αφρικανική Ήπειρο. Έχουμε λοιπόν τρία επίπεδα. Το διαπροσωπικό επίπεδο, ε, το επίπεδο μεταξύ επιχειρήσεων και βέβαια τις διακυβερνητικές σχέσεις. γιατί βεβαίως ε, υπάρχει αυτή η εδαφική στρατηγική ανάπτυξης για δημιουργία εισοδήματο, ε, η αηφόρος διαχείριση φυσικών πόρων και η κλιματική δράση, αηφόρος μετασχηματισμός της Αφρικανικής Γεωργίας ε, και η ανάπτυξη της αγοράς εργασίας. Αυτό βεβαίως ε, περιλαμβάνεται και στο βασικό μας πρόγραμμα, το λεγόμενο ΚΑΝΤΕΠ, το συνολικό πρόγραμμα για την γεωργία στην Αφρική, ε, το οποίο είναι το πρόγραμμα για το 2063, το λεγόμενο «Η Αφρική που θέλουμε». Και βεβαίως ε, η ομάδα αυτή εργασίας πρότεινε και κάποιες άλλες συστάσεις Οπότε... Χαίρομαι για το ότι μας δώσατε την ευκαιρία να έρθουμε εδώ πέρα και να μοιραστούμε την έκθεση αυτή μαζί σας και ελπίζω να μπορέσουμε έτσι να μετασχηματίσουμε την γεωργία στην Αφρική για να σταματήσει η πείνα, να τελειώσει η πείνα μέχρι το 2025. Αυτό είναι άλλο από την Ατζέντα 2030 που όπως ξέρετε έχει στόχο το 2030. Εμείς έχουμε στόχο το 2025 γιατί θεωρούμε ότι η πείνα είναι ένα βασικό ζήτημα και βεβαίως ε, και ο υποσυτισμός είναι σοβαρό θέμα στην Αφρική. Πρέπει να επιταχύνουμε να υπάρξει κάποια πρόοδο πρόοδο, με συγχωρείτε, Προσπαθούμε λοιπόν να εφαρμόσουμε τις ευρύτατες αυτές συστάσεις ε, για να μπορέσουμε να βασιστούμε και στην υφιστάμενη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικανικής Ένωσης στον ευρύτερο τομέα των τροφίμων και της ε, γεωργίας για να επιταχύνουμε την αηφόρο ανάπτυξη του τομέα αυτού στην Αφρική και βεβαίως να εστιάσουμε ειδικά στο πώς θα υποστηρίξουμε καλύτερα τους νέους και τις ε, γυναίκες. Κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτές, ε, βασίζομαι στην στήριξή σας ε, για το πρόγραμμα αυτό και ελπίζω να επανέλθω για να σας ενημερώσω για την πρόοδο του πολύ σημαντικού αυτού προγράμματος. Σας ευχαριστώ, μούτσας γκράσιας και μερσί μποκού και σούκρεμ. Σας ευχαριστούμε κυρία Σάκο για την προθυμία σας και το πόσο διαθέσιμοι είστε να έρθετε στην Επιτροπή. Περνάμε στην Ομιγύρη. Χρόνο έχουμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να μακρηγορούμε. Έχουμε πάντως αρκετό χρόνο για να λάβουν το λόγο στο ζήτησαν. Η κυρία Σρέιρ πρώτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι είμαι υπερήφανη για το ότι ε, είμαι παρούσα αυτήν την στιγμή. Συχνά στην Ευρώπη μιλάμε για τα προβλήματα του ασύλου και τέτοια θέματα και αυτήν την στιγμή έχουμε μια πολύ καλή παρουσίαση για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την ε, Αφρική. Είμαι και στην αντιπροσωπεία για την ε, Αφρική. Είμαι λοιπόν υπερήφανος για την Ευρώπη και για τον Επίτροπο για την πρόταση αυτή και νομίζω ότι πρέπει πραγματικά να βοηθήσουμε και με τους κορυφαίους επιχειρηματίες και οπωσδήποτε έχει εμπλακεί σχετικά η Ολλανδία. Θα ήθελα να φέρω κάποια πραγματάκια. Παρατηρούμε σε πάρα πολλά προγράμματα για την Αφρική ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μιλάνε, πίνουν, τρώνε, παίρνουν τις ε, πτήσεις ε, first class, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο. Οπότε το ζήτημα είναι ακριβώς ε, να έρθουν και οι αγρότες και να υπάρχουν άμεσες επαφές με τους ενδιαφερόμενους και όχι τόσα πολλά πέρα δόθηκε. Μια που μιλάμε για την ισότητα των φύλων, επίσης βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Ε, κοιτάξτε, και εσείς και εγώ γυναίκες είμαστε, μπορούμε να τα δούμε πιο άμεσα αυτά τα ζητήματα σε μια απευθείας ε, επαφή. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να εμπλακούν και οι οργανώσεις των αγροτών, κόπα, κοζέκα και βεβαίως και το εμπόριο των αφρικανικών χωρών μεταξύ τους είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει πολύ και βεβαίως το σημαντικότερο το οποίο είπα πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους Αφρικανούς ε, γεωργούς ε, ε, γελάνε λίγο οι συνάδελφοι για να μπορέσουν ε, να λάβουν μέρος ε, και να ανταποκριθούν στις διεθνείς ποιοτικέ απαιτήσει. Ακριβώς θα πρέπει να ε, ανταποκριθούν. Να βοηθήσουμε λοιπόν την Αφρική, να μην φεύγει ο κόσμος από εκεί. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για το ότι είστε εδώ αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς πρέπει να φύγω τώρα για να πάω σε μια άλλη συνεδρία. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και ε, οι βοηθοί μου εδώ πέρα θα μεταφέρουν το όσο θα πείτε. Σας ευχαριστούμε κυρία Σρέιερ. Κυρία Χόιμπουχ. Ja, herzlichen Dank, herzlichen Dank. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ξανά ήρθατε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι μας μεταφέρατε την άποψη της Αφρικανικής Ένωσης και την Κομισιόν της Αφρικανικής ε, mm-hmm. Ένωσης. Εγώ βρίσκομαι και στην Επιτροπή Ανάπτυξης, είμαι μέλος και χαίρομαι. Ακριβώς για τον συντονισμό που έχουμε, εσείς ε, αυτή τη στιγμή αναπτύσσετε μια κοινή στρατηγική για ολόκληρη την Αφρικανική Ήπειρο. Ακριβώς τονίστηκε ότι οι νέοι χρειάζονται δουλειά και εκεί πέρα οι γεωργοί παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτή την εβδομάδα ε, οργάνωσα με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων μια διάσκεψη για την καταπολέμηση της ε, πείνας και ακριβώ αυτό το οποίο ακούστηκε ήταν ότι σημαντικές είναι οι μικρές επιχειρήσεις. Ε, εκεί πέρα μπορεί να καταπολεμήσουμε την πείνα, να υπάρξει μια τοπική οικονομία και για την πρόσβαση στην, ε, στις αγορές ε, και βεβαίως εδώ πέρα σκεφτόμαστε κυρίως την ευρωπαϊκή αγορά αλλά πρέπει να δούμε και την αφρικανική αγορά ως εσωτερικό εμπόριο το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί και εδώ πέρα και ο Επίτροπος Χόγκαν και εσείς αναφέρατε την συνοχή της ε, πολιτικής και τα έχουμε πει δίμερος υπάρχει ένα μικρό κομμάτι για την ε, συνοχή της πολιτικής στην ανακοίνωση της ε, Κομισιόν. Η, ανάπτυξη, η Επιτροπή Ανάπτυξης ε, έχει βγάλει μια γνωμοδότηση όπου πάλι τονίζει ότι πρέπει να έχει μια συνοχή η πολιτική μας και στην μεταρρύθμιση της γεωργίας και να συνδεθούν τα διάφορα αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω κύριε Χόγκεν να μας στηρίξετε και στον τριμερή διάλογο γιατί είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά αναγκαίο. Αν συντονιστούμε λοιπόν και έχουμε μια κοινή στρατηγική, θα ασκήσουμε μια συνεκτική ε, πολιτική. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει ειδικά στον τομέα των Υπουργών ε, Γεωργίας ε, και να δούμε το τι επιδράσεις έχει, το τι κάνουμε εδώ πέρα σε αγορές σε άλλα μέρη του πλανήτη. Αυτό πρέπει να μπει στην μεταρρύθμιση της ε, γεωργικής πολιτικής. Τώρα, προς την ε, μεριά του Συμβουλίου θα έπρεπε να μιλήσουμε όχι μόνο με τους Υπουργούς ε, Γεωργίας αλλά και με τους Υπουργούς Αναπτυξιακής Βοήθειας για να ρίξουν μια ματιά στο θέμα. Και έτσι νομίζω θα προχωρήσουμε κάπως. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μαγκίνες έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Ε, κύριε Σάκο, εκτιμούμε ιδιαίτερο τη δική σας παρουσία και φυσικά Τιμ Άρνολτ, εκτιμούμε ιδιαίτερο και αναγνωρίζουμε το δικό σας έργο. Και ε, χαιρόμαστε και για την ε, ανάμειξη και τη δέσμευση του κυρίου Χόκου, του επιτρόπου μας για το θέμα αυτό. Όταν το πρόβλημα είναι τεράστια, ε, πολλές φορές προτιμούμε να εθελοτυφλούμε και αυτός ο αριθμός των 800 εκατομμύρια έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Δεν μπορούμε να ε, εθελοτυφλούμε απέναντι στα προβλήματα. Είναι θέματα που ενδιαφέρουν και το δικό μας μέλλον και το μέλλον της Αφρικής και έχουμε ένα ηθικό, διοντολογικό καθήκον να εμπλακούμε στην ανάπτυξη της Αφρικής, αλλά είναι και προς το συμφέρον μας να μεριμνήσουμε για τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και τη δημιουργία ευκαιριών στην Αφρική και μια και ο Επίτροπος, ο Τόμαν και εγώ είμαστε από μια χώρα που έχει βιώσει ε, το λοιμό και εκατοντάδες ε, εκατομμύρια χρειάστηκε να αποδημήσουν ή πολλοί συμπολίτε μας έχασαν τη ζωή ε, του λοιμού. βλέπουμε πόση πιθανότητα υπάρχει και δυνατότητα για βελτίωση και ανάπτυξη της γεωργίας. Είμαστε ζωντανοί μάρτυρες και απόδειξη αυτών. Τι συγκεκριμένη συνεισφορά μπορούμε να πραγματοποιήσουμε για την αγροτική ανάπτυξη της Αφρικής. Ευχαριστώ και χαίρομαι ιδιαίτερως για την παρουσία σας εδώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Χόισλινγκ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ και για την ε, παρουσίασή σας. Αυτό το οποίο μας είπατε. Παρ' όλα αυτά ε, προκύπτουν κάποια ερωτήματα. Έφυγε η κυρία Σράιερ τώρα και είναι ζητήματα κυρίως εμπορικής πολιτικής. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι το θέμα δεν είναι η Ευρώπη να έχει ανοιχτές Αφρικές και η Αφρική κλειστές αγορές και να υποφέρει έτσι η Αφρική για το ότι ε, αναγκάστηκαν τελικά να ανοίξουν τις ε, αγορές τους ε, και να έρχονται ευρωπαϊκά προϊόντα σε τιμές σε οποίες δεν μπορούν να παράγουν η αφρικανή παραγωγή. Εμείς επιδοτούμε πολλά λεφτά κάθε χρόνο την γεωργία μας, αλλά δεν είναι δυνατόν δηλαδή να καλλιεργούμε προϊόντα στην Αφρική συχνά μετανάστες και να τα εξάγουμε μετά στην ε, Αφρική. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα όσο και αν δεν θέμε να το ακούμε στην Αύρη, θεωρούμε εμείς την Αφρική έναν τρόπο και ένα μέρος εξαγωγής των πλεονασμάτων μας. Είτε μιλάμε για προϊόντα γαλαξιού, είτε για οτιδήποτε άλλο. Και τώρα προσπαθούμε το αντίθετο να το φορολογήσουμε. Μπορεί να λειτουργήσει κάτι τέτοιο και να λέμε «Α, ναι, τώρα μάθετε εσείς από εμά, θα σας δώσουμε λεφτά για την ανάπτυξη». Και Φοβάμαι ότι τα πράγματα θα γίνουν όπως και σε πάρα πολλά άλλα έργα, δηλαδή να παράγονται προϊόντα για να εξάγονται στις ευρωπαϊκές αγορές. Είχε προϋποστηρίξει διάφορα προγράμματα, ας πούμε, παρόμοια η Γερμανία, για να εξάγεται ε, ζάχαρη στην Ευρώπη και να μην ε, μένει η παραγωγή στην, ε, στον τόπο. Πρέπει λοιπόν ε, η Αφρική να αναπτύξει το δικό της αγροτικό μοντέλο. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμεί εξαγωγή του δικού μας ε, μοντέλου, της υψηλής τεχνολογίας, της εντατικής καλλιέργειας. Πρέπει να βρει τον δικό της ε, το δρόμο η Αφρική και εμείς να την στηρίξουμε. Δεν ξέρω, εκτός αν θέλετε να αντιγράψετε κάτι το έτοιμο. Υπάρχουν προβλήματα βεβαίως, η Αφρική χρειάζεται και δικές τιμές για τα ε, προϊόντα Βλέπουμε και στο κακάο και στον καφέ υπάρχει dumping τιμών από την Ευρώπη ε, και δεν έχουν καμία ευκαιρία η παραγωγή. Θα πρέπει λοιπόν οι εισαγωγές ε, να πληρώνουν σωστές τιμές για να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Και αυτό νομίζω θα έχει καλύτερα αποτελέσματα από το να δώσουμε λεφτά έτσι, Εντάξει, δίνουμε λεφτά για να έχουμε καλή ισχύ τη συνείδησή μα, αλλά τελικά δεν λύνεται το πρόβλημα. Ευχαριστούμε κύριε Χόισλινγκ. Και τελευταίο μιλητή ο κύριο Φλάναγκαν. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσε η παρουσιάσει και από του τρει καλεσμένου μα. Και χαίρομαι που ξαναβλέπουμε το μετά την τελευταία φορά, τελευταία συνεδρίαση. Σε όλη μου τη ζωή, δεν είμαι και πολύ μεγάλο, είμαι 47 ετών, σε όλη μου τη ζωή έγινα μάρτυρα καταστάσεων όπου κάναμε έρανο και συγκεντρώναμε χρήματα για να βοηθήσουμε την Αφρική. Ακόμη και στο σχολείο όταν πήγαινα ε, κάναμε εράνους για την Αφρική και στη γειτονιά μου. Ε, πάντως θυμάμαι έπαιξα έπαιζα γκολφ για 15 ώρες ε, συνεχόμενες ε, για να μαζέψω χρήματα για την Αφρική. Και όταν είχαμε το λοιμό στην Αιθιοπία, επίσης ε, κάναμε ράνους. Ήμουν πολύ νέος τότε, πολύ μικρός. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να βοηθήσουμε. Γιατί σκεφτόμουν ότι θέλω να βοηθήσω γιατί και εγώ αν πεινούσα και τα αδέρφια μου πεινούσαν θέλει κάποιος να με βοηθήσει. Πάντω ε, μετά που συγκεντρώσαμε τα χρήματα και τα στείλαμε στην Αφρική, διαπιστώσαμε ότι τότε η Αιθιοπία εξήγαγε ε, σιτηρά. Ενώ οι κάτοικοι λιμοκτονούσαν. Και μάλιστα και το, η επιχείρηση McDonald's συμμετείχε και μάθαμε ότι γινόταν εξαγωγές τροφίμων τη στιγμή που ο πληθυσμός λιμοκτονούσε. Το ίδιο και στην Ιρλανδία. Μερικοί ε, το αποκάλεσαν λιμό, άλλοι γενοκτονία. Δεν μ' αρέσει ε, όρος πλημμύρα ε, να χρησιμοποιείται για τους 160.000 ε, Ιρλανδούς που μέσα σε δύο-τρεις εβδομάδες έφτασαν στο Λίβερμπουλ. Μερικοί το ε, χαρακτήρισαν ως μεταναστευτική πλημμυρίδα. Δεν μ' αρέσουν αυτοί οι ορισμοί για τα μεταναστευτικά κείμενα. Ήταν άνθρωποι που προσπάθησαν να ξεφύγουν από το λοιμό τότε από την Ιρλανδία. Και όταν οι άνθρωποι λιμοκτονούν, παρόλα αυτά υπάρχουν κυβερνήσεις που θεωρούν δεν έχουν ε, επιλογή γιατί είναι τόσο υπερχρεωμένες, ίσως μερικές φορές παρά είναι έντιμες και παρόλα αυτά συνεχίζουν να εξάγουν τρόφιμα ενώ ο λαός τους λιμοκτονεί. Λυπάμαι αν είναι άσχετο αυτό που λέω, αλλά αφορά κάτι με τα, τα τρόφιμα που καταναλώνουμε και εδώ και στην Αφρική, κυρίως τα, τα ψάρια. Άκουσα πολλές και διάφορες ιστορίες, δεν ξέρω αν αληθεύουν ή όχι. Η, η σούπερ τράτα, σούπερ μηχανότρατα είναι μια ιστορία που ακούμε. Ακούμε τέτοιες τεράστιες μηχανότρατες που αλλιεύουν στις ακτές Αφρικής, μάλιστα εκεί ξεχωρικά υδάτα που γινόταν παραδοσιακή αλία για εκατοντάδες χρόνια και τώρα έχουν ε, εξολοθρευτεί τα ηχθιαποθέματα. Μπορεί κάτι να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφύγει τέτοια βιομηχανική αλία. Επίσης αναφέρθηκε η κοινή γεωργική πολιτική και η μεταρρύθμισή της. Στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει και την κατάσταση στην Αφρική. Ακούσαμε τον Επίτροπο Χόγκαν που είναι και συμπατριώτης μου και ότι μάλλον το ίδιο. Ακούσαμε τα, τη φρίκη του λίμου Υπάρχει κάτι όμως που μπορούμε να κάνουμε στην ΚΑΠ και για την Αλία το ίδιο για να βελτιωθεί η κατάσταση. Επίσης την κυρία Σάκο που έκανε τον κόπο και έκανε αυτό το μεγάλο ταξίδι για να έρθει εδώ σήμερα την ευχαριστούμε γιατί μίλησε πολύ σωστά. Και τελευταίο αυτή τη φορά όντω τελευταίο ο ο κύριο Σεχάου Σάντο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τους καλεσμένου μα τον κύριο Τόμ Άρνολτ, τον Επίτροπο Φιλ Χόγκαν και την Επίτροπο Γιουζέφα Σάκο, που κατάγεται από την Αγκόλα και άρα έχουμε και κοινή γλώσσα. Και θα ήθελα να εξάρω το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη συνεργασία με την Νέα Αφρική. Ε, μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν από τους βασικούς δωρητές στην Αφρική και χώρες που περισσότερο συνεργάστηκαν με την Αφρική. Και εγώ για την Αλία θα ήθελα να μιλήσω, με πρόλαβε μάλιστα ο Ιρλανδός συνάδελφος. Εγώ συμμετέχω και στην ΑΚΕ Ασχολήθηκα πολύ με την Αφρική και κυρίω με τα θέματα της ε, θάλασσας, ε, ε, της αλίας, της γεωργίας και γενικώ με το θέμα των, της αγροτικής οικονομίας, της, των γεωργικών τροφίμων, της αλίας αλλά και της ηχθειοκαλλιέργειας, της ηχθειοτροφίας. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες εκεί στην Αφρική. Έχουμε στην κοινή αλληλευτική μας πολιτική αλληλευτικές συμφωνίες για βιώσιμη αλεία. Και Μάλιστα, ήμασταν πολύ διαφορετική συμπεριφορά μας απέναντι στην παράνομη αελία από ό,τι άλλες περιοχές του κόσμου. Και μάλιστα στις Βαχάμες πριν από δύο χρόνια υπολογίστηκε ότι οι ζημίες από άναρχη και παράνομη αλία είναι τεράστιες, δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι οι ζημίες από την παράνομη άναρχη και αδήλωτη αλία στις ε, αφρικανικές χώρες. Από αυτά που άκουσα από τον κύριο Τόμ Άρνολτ μου δημιουργήθηκε ένας προβληματισμός. Δεν αναφέρθηκε μια άλλη πολύ σημαντική χώρα στην περιοχή, η Κίνα. Γιατί η Κίνα είναι μια πολύ ε, σημαντική δύναμη και πολύ σημαντικός παράγοντας αυτή της κακέρα της Αφρικής. Και μεταξύ άλλων η Κίνα προωθεί μια συνεργασία και γεωργική με την Αφρική, συνάπτοντας πολλές συμφωνίες με πολλές αφρικανικές χώρες. Ε, σε 33 χώρες, 744 γεωργικές συμφωνίες έχει συνάψει η Κίνα, με τη Μοζαμβίκη για παράδειγμα. Ε, έχει συνάψει συμφωνία 700.000 ε, ευρώ για νέες γεωργικές υποδομές. Και στην ΑΚΕ διαπιστώσαμε ότι στο διάλογο με την Αφρική το θέμα της Κίνας είναι αρκετά λεπτό και δύσκολο. Το διαπιστώσαμε αυτό επανειλημμένος. Ένα από τα ζητήματα είναι το πολιτικό. Ε, στην σχέση μας με την Αφρική, η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει πολλούς όρους. Σε αντίθεση με την Κίνα που δεν εφαρμόζει καμία αιρεσιμότητα, δεν βάζει καθόλου όρους στη συνεργασία της με την Αφρική. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Οπότε σε αυτό το σχέδιο δράσης που έχουμε για την ανάπτυξη της διατροφής της υγείας στην Αφρική, πώς λαμβάνουμε υπόψη το ρόλο της Κίνας. Γιατί η Κίνα δεν είναι άσχετος παράγοντας, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στον κόσμο και ιδιαίτερα στην Αφρική. Πώς λαμβάνετε υπόψη το ρόλο της Κίνας, τη θέση της Κίνας και πώς βλέπετε το μελλοντικό ρόλο και παρουσία της Κίνας στην Αφρική. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Σεράο Σάντος. Δεν ζήτησε άλλο συνάδελφος το λόγο. Α, και κάτι άλλο. Σας ζητώ συγγνώμη. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να μείνω μέχρι το τέλος. Αλλά επειδή είμαι πρόεδρος σε ένα σεμινάριο που συμπίπτει, μη με κακοκάρδεις, μην ε, με παρεξηγήσετε αν χρειαστεί να φύγω πριν το τέλος συνεδρίας, αλλά πρέπει να προεδρεύσω στο workshop. Ναι, όντως, γνωρίζω σε Ξέρω ότι σε λίγα λεπτά πρέπει να φύγεις γιατί θα προεδρεύσεις στο σημαντικό αυτό workshop, ε, Ρικάρδο. Μην ανησυχείς λοιπόν. Και για να ολοκληρώσουμε θα δώσω το λόγο και πάλι στους καλεσμένους μας. Πρώτα στον κύριο Τόμ Άρνολτ και μετά στους επιτρόπους. Θα ήθελα να μας σχολιάσετε αυτά που ακούσατε από τη συζήτηση. Για να ολοκληρώσουμε. Έχετε το λόγο κύριε Άρνολτ. Yeah, thank you very much Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αρκετά από αυτά τα σχόλια. Κάποια φράση χρησιμοποιήθηκε. Περί οικονομικής ζωτικότητας και θέσεων εργασίας. Και κατά κάποιο τρόπο αυτή είναι η καρδιά του θέματος. Στο επίκεντρο αυτό που συστήνουμε, κυρίως την εδαφική προσέγγιση για την απασχόληση. Όλοι γνωρίζουμε, το ξέρουμε και από την Ευρώπη αλλά και από αλλού, ότι ο καλύτερος τρόπος να εγγυηθεί κανείς ότι πολλοί άνθρωποι μπορούν να ασχολούνται με τη γεωργία είναι να τους δώσει περισσότερες ευκαιρίες για να έχουν εισόδημα και εκτός γεωργίας. Αυτό είναι το υπόβαθρο που μας οδήγησε στο να συστήσουμε εδαφική προσέγγιση. Παραδεχόμαστε ότι στο σχεδιασμό για το μέλλον η Αφρική πρέπει να επενδύσει στην οικονομική ζωτικότητα της υπαίθρου. Εν μέρη αυτό σημαίνει επενδύσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε μεσαίου μεγέθους πόλεις. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Μπορούμε να βελτιώσουμε την ε, παραγωγικότητα και την οικονομική βιωσιμότητα των γεωργών. Σε κάθε περίπτωση αυτό μπορούμε να το βοηθήσουμε αν καταστήσουμε την οικονομία της υπαίθρου πιο ζωτική, πιο ε, ζωήρη αν θέλετε. Αναφέρθηκε και το εμπόριο. Ποια είναι η αφετηρία μας. Ότι η αφρικανική αγορά τροφίμων ε, επεκτείνεται τάχιστα. Λόγω αυξήσεως του πληθυσμού και λόγω αυξανωμένης μεσαίας τάξης. Άρα αυξάνεται η ζήτηση για τρόφιμα διαφόρων ειδών. Μέχρι τώρα σημαντικό ποσοστό της αυξημένης ζήτησης εκαλύπτεται από εισαγωγές από χώρες εκτός Αφρικής. Τι λέμε εμείς. Ότι ο αφρικανικός τομέας των τροφίμων έχει μια πραγματική ευκαιρία τα επόμενα 10-15 χρόνια να μπορεί να καλύπτει την εσωτερική ζήτηση. Για να το πετύχει αυτό όμως θα πρέπει να αλλάξει η βιομηχανία τροφίμων τη Αφρικής. Σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι καν ανταγωνιστικός ο τομέας εν σχέση με τις εισαγωγέ. Χρειάζεται επενδύσει, να αυξηθεί η δυνατότητα να προσθέτει αξία στην αφρικανική παραγωγή. Και υπάρχουν και πραγματικά σημαντικά ζητήματα για πρότυπα ασφαλείας τροφίμων και υγειονομικά και φυτο πρότυπα και προδιαγραφές. Πρέπει να βελτιωθούν σε πάρα χώρες. Και τι λέμε εμείς, ότι υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία για δομημένη και βιώσιμη συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. Συνεργασίας για τη βελτίωση αυτών των προδιαγραφών. Αν περί αυτού πρόκειται, τότε έχουμε τα θεμέλια για την αύξηση ενδοαφρικανικών συναλλαγών και εμπορίου. Σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να είναι το εμπόριο, ε, είναι ελάχιστα ανεπτυγμένο. Και η Αφρικανική Ένωση ίδια τον αναγνωρίζει και λέγει ότι θέλει να αυξηθεί το ενδοαφρικανικό εμπόριο. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πρέπει να αντιμετωπιστούν κάποια από τα υποκείμενα προβλήματα. Έλλειψη ανταγωνιστικότητα, η ανάγκη βελτιώσεω της ασφαλεία των προδιαγραφών ασφαλεία τροφίμων και συμμόρφωση με πρότυπα SPS. Εάν γίνουν αυτά, δεν μιλάμε τώρα για βραχυπρόθεσμες λύσεις, αλλά μακροπρόθεσμο όραμα βελτιώσεων και προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή θα είναι η βάση όχι μόνο για βελτίωση ενδοαφρικανικού εμπορίου, αλλά να αυξηθεί και η δυνατότητα Αφρικής να μπορεί να εμπορεύεται διεθνώς. Οπότε ερχόμαστε σε κάποιες από και τα σχόλια που ακούστηκαν. για τις παρούσες εμπορικές ε, πρακτικές και το dumping. Το αντιμετωπίζουμε αυτό στην έκθεσή μας, το βαθμό που ιχνηλατούμε τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η εμπορική ε, πολιτική τις τελευταίες δεκαετίες. Τι λέμε. Ότι είναι πολύ διαφορετική πολιτική σήμερα αν συγκρίσουμε πριν από 20-30 χρόνια. Δύσκολο λοιπόν να αρνηθούμε ότι οι μηχανισμοί που είχε θεσπίσει η Ευρώπη όπως εξαγωγικές επιστροφές οδηγούσαν άμεσα σε dumping στις αφρικανικές αγορές και ήταν επιζήμιες. Αυτές οι βασικές διεθετήσεις έχουν μεταλλαχθεί, έχουν αλλάξει. Δεν υφίστανται πλέον οι εξαγωγικές επιστροφές. Έχουν σταματήσει από τον Ιανουάριο του 2016. Επίσης, υπήρξε και αλλαγή όσον αφορά την πολιτική για την ανάπτυξη που λαμβάνεται όλο και πιο σοβαρά υπόψη. Χρειάζεται λοιπόν συνεχτική πολιτική για την ανάπτυξη. Δηλαδή, τι σημαίνει διασύνδεση μεταξύ αγροτικής πολιτικής, αναπτυξιακής πολιτικής, περιβαλλοντικής πολιτικής, εμπορικής πολιτικής. Παραδεχόμαστε ότι πιθανότατα περισσότερα μπορούν να γίνουν σχετικά με όλα αυτά. Και έχουμε συστήσει κάποια πράγματα και σαν τμήμα της διαδικασίας που ακολουθήσαμε διαβουλευτήκαμε με ενδιαφερόμενους φορείς στην Ευρώπη και στην Αφρική να το συζητήσουμε αυτό και ο Επίτροπος όπως είπε θεωρεί ότι πρέπει να τονίσουμε περισσότερα τα θέματα αυτά. Επουδενή δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει τελειώσει το θέμα αλλά είμαστε διαφορετική θέση τώρα από ό,τι πριν από 10-20 χρόνια. Ερχόμενος τώρα σε κάτι άλλο, χωρίς να επισέλθω σε λεπτομέρειες, σε αυτό που ανέφερε ο Μικ Φλάναγκαν, αναφέρθηκε σε κάποια σημαντικά ζητήματα. Αυτό πιστεύω. Λέμε στην έκθεση ότι υπάρχουν κάποια θέματα που θίγουμε όσον αφορά τη διακυβέρνηση. Η διακυβέρνηση σαν υπόβαθρο. Η βελτίωση της διακυβέρνησης στην Ευρώπη, στη γνώμη στην Αφρική, θεωρείται ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη. Και η Αφρική προδεύει εν γέννη. Αλλά υπάρχουν κάποιες αφρικανικές χώρες που ακόμα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διακυβέρνησης και σε κάποιες περιπτώσεις αυτό αντικατοπτρίζεται σε συγκρούσεις και σειράξεις. Ο αριθμός αφρικανικών χωρών που βρίσκονται σε συγκρούσεις ή παρατεταμένη κρίση όπως αποκαλείται είναι σημαντικός. Το λέμε αυτό για να τονίσουμε πραγματικά ότι αν θέλουμε να πετύχουμε ανάπτυξη και πιο συγκεκριμένα να πετύχουμε βελτιώσεις στον αγροτροφομικό τομέα και στην οικονομία της υπαίθρου, το υποκείμενο πρόβλημα της αντιμετωπίσεως των συγκρούσεων ε, πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και αυτή είναι μια πρόκληση για την Αφρική μια πρόκληση για τη διεθνή κοινότητα. Δεν θα εκπλήσει κανένα ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ζήτησε αυτό που αποκάλεσε μια, ένα κύμα διπλωματίας για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, να, προληφθεί, να προληφθούν οι κρίσεις και να επιληθούν οι κρίσεις. Και θεμελιωδώς αυτό θα πρέπει να γίνει εάν θέλουμε να υπάρξουν συνθήκες για ανάπτυξη της Αφρικής. Και έχουμε τη σύγκρουση σοβαρά προβλήματα περί ασφαλείας τροφίμων και σε σπάνιες περιπτώσεις έχουμε λοιμό. Τα στατιστικά μας δείχνουν ότι από το 2014 μέχρι το 2017 ο αριθμός ανθρώπων στην Αφρική που υποφέρει από σοβαρή ε, ανασφάλεια τροφίμων, έλλειψη τροφίμων από τα 260 εκατομμύρια έφτασε τα 375 εκατομμύρια. Και βασική εξήγηση γι' αυτό είναι οι συγκρούσεις αντιμετώπιση αυτών των υποκειμένων προβλημάτων είναι θεμελιώδου σημασίας για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία που θέλουμε. Τι συζητάμε. Συζητάμε ιδέες που μπορούν να εφαρμοστούν με τον καλύτερο τρόπο σε ένα σταθερό πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον και δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα σε όλες τις αφρικανικές χώρες. Αυτό που δεν, δεν ισχύει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο Επίτροπος Χόγκαν έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εν συντομία να προσθέσω και εγώ κάποια στις πλήρεις απαντήσεις που έδωσε ο Τόμας. Η Αφρική πρέπει να δώσει, να ηγηθεί πολιτικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δώσει τεχνογνωσία, εμπειρία και οικονομική υποστήριξη. Αυτή είναι η διαφορά. Η Αφρική πρέπει να ηγηθεί. Δεν θα επιφέρουμε διαφορετικά τις ε, βελτιώσεις που θέλουμε στην Ήπεθρο και στη Γεωργία που θα παίξει ρόλο για να πετύχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ανθρώπους, για τους λαούς της Αφρικής, τον αυξανόμενο πληθυσμό της ε, Αφρικής. Αυτή η έκθεση λοιπόν στο πνεύμα συνέχιση του διαλόγου θέλει διαβουλεύσει από τώρα μέχρι τον Ιούνιο. Θέλουμε διαβουλεύσει από τώρα μέχρι τον Ιούνιο για την έκθεση. Να τοποθετηθούν οι διάφοροι. Να πούν αν διαφωνούν, αν θέλουν βελτιώσει σε την έκθεση. και α και εγώ. Θα συναντηθούμε στη Ρώμη τον Ιούνιο. Έχουμε διπουργική συνάντηση που θα δράζεται από τις διαβουλεύσεις να δούμε πώς θα εφαρμόσουμε τα πορίσματα και τις ε, κατευθύνσεις εκθέσει. Έχουν πολλέ εκθέσει και το σημαντικότερο όμω είναι πώ να εφαρμόσουμε αυτά που λένε οι εκθέσεις. Αναφέρθηκα βραχυπρόθεσμη στόχοι. Έχουμε μεσομακροπρόθεσμες ε, προσεγγίσεις. Θα πρέπει να υπάρξει μια μάθα δημιουργηθεί και ένα σχέδιο εφαρμογής. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό θα το κάνουμε στη Ρώμη. Να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Μάμιτσα και τους ανθρώπους της ΔΕΦΚΟ, τον Επίτροπο Μίμιτσα και τους ε, ανθρώπους της ΔΕΦΚΟ που βοήθησαν, όπως και οι δικοί μου της DG Agri με βοήθησαν και η ομάδα του Tom Ireland βοήθησαν να συντάξουμε και να παρουσιάσουμε αυτή την έκθεση. Πολλέ παραπομπέ στην έκθεση υπάρχουν και αναφορέ, αν τη διαβάσετε μετά από σήμερα, που αναφέρεται στην συνεκτική πολιτική. Ήταν επικοδομητικέ συζητήσει που έγιναν. Μαρτιν, ήσουν πολύ αρνητικό μα αυτά. Και τα και εγώ είχαμε πολύ καλύτερη συνεννόηση. Κεφάλαιο 6-4. Βοηθάει με στοιχεία και όπως είπε και ο Τόμας, πρέπει να παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα. Να ξέρουμε ότι αυτό που εξάγεται δεν είναι στην περίπτωση των προϊόντων των ε, ευρωπαϊκών που γίνονται, που τα, τα ρίχνουμε στην Αφρική. 3,7 δισεκατομμύρια εμπόριο έχουμε από την Αφρική προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αμφίδρομη η διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί. Πρέπει να υπάρχουν ισότιμε συνθήκε που επικρατούν. Δίνουμε προτιμησιακή ε, ε, προσέγγιση στην Αφρικανική Ένωση, στι χώρε Αφρικανική Ενώσεω, όσον αφορά δασμού και ποσοστώσει για διάφορα προϊόντα. Έχουμε εξαλείψει επί την ηγεσία τη δική μου τη κυρία Μάλστρομ στο Ναϊρόμπι του 2015 όλε τι επιδοτήσει που στρεβλώνουν την αγορά, την εμπορική. Αυτό δεν το αναφέρατε, αλλά αυτό συνέβη και άρα έχουμε μεγάλες βελτιώσεις. Και βεβαίως συμφωνώ δεν είναι τα πάντα τέλεια αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να αλλάζουμε την πολιτική και να τη βελτιώνουμε. Και σίγουρα θα λαμβάνω υπόψη το στοιχείο της συνοχής πολιτικής και της μεταρρυθμίσεως της ΚΑΠ. Η κυρία Μαγκίνης έχει απόλυτο δίκιο. Αυτά τα αποτελέσματα έχουν σημασία. Μπορεί να γράφουμε όσοι εκθέσεις θέλουμε, αλλά πρέπει να δώσουμε αποτελέσματα. Και αυτό που κάνουμε είναι να δώσουμε την τεχνογνωσία μας, την οικονομική μας υποστήριξη Είμαστε ο μεγαλύτερο δοτή τη Αφρική. Όπω είπε ο κ. Φλάνακα, θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι πηγαίνουν στο σωστό στόχο, στου σωστού ανθρώπου τα χρήματα. Να μην μπλέκονται διάφοροι ε, ενδιάμεση. Θέλουμε τελικά να πετύχουμε τα αποτελέσματα για το, για το λαό που θέλουμε. Λοιπόν, έχουμε ιστορικό κοινό, ιστορικό σαν Ιρλανδοί, ε, και είμαστε ένα είδος ε, ιεραπόστολοι στη δουλειά που κάναμε. Έχουμε κοινέ αξίες με τον κύριο Φλάνναγκαν. Με εκπλήσει που είχατε χρόνο να παίξετε γκολφ. Με εκπλήσει που είχατε χρόνο να παίξετε γκολφ. Ε, δεν το πίστευα αυτό. Έχετε και ελεύθερο χρόνο. Μπράβο. Για αναψυχή. Ε, όχι για μερικούς μήνες ακόμα τον Ιούνιο θα δείτε τι, αν μπορείτε να πετύχετε αναψυχή ε, μέσω του γκολφ. Ο κ. Σάντσετς μια ερώτηση προς την κυρία Σάκο όσον αφορά την Κίνα ε, και θα, θα αφήσω την κυρία Σάκο να απαντήσει για το θέμα της ε, Κίνας. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Και η τελευταία η Επίτροπος η κυρία Σάκο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά το ενδοαφρικανικό εμπόριο. Με αυτό θα ξεκινήσω. Γιατί ε, αναφέρθηκε από πολλούς την ε, αύξηση του ενδοαφρικανικού εμπορίου. Πέρυσι το Μάρτιο εμ, εγκαινιάσαμε την ζώνη ελεύθερου εμπορίου στην Αφρική. Έγινε στο Κιγκάλι αυτή η επίσημη έναρξη και θέλουμε τώρα να περάσουμε στην υλοποίηση αυτού του χώρου ελεύθερου εμπορίου. Συνεργαζόμαστε με τη ΦΑΟ, το Παγκόσμιο Οργάνωση Εμπορίου ε, και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και θα έχουμε και την πρώτη διεθνή διάσκεψη για την ασφάλεια των τροφίμων, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Αν θέλουμε εμπόριο, θα πρέπει να παράγουμε ποιοτικά προϊόντα, είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο και θα πρέπει να πληρούμε όλες τις προδιαγραφές της ασφάλειας των τροφίμων. Το περασμένο μήνα, το Φεβρουάριο, οργανώσαμε λοιπόν την πρώτη διεθνή διάσκεψη για την ασφάλεια των τροφίμων. Και μάλιστα εκεί συμμετείχε η Αφρικανική Ένωση, η ΦΑΟ και η Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου. Μάλλον η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Έγινε στην έδρα της Αφρικανικής Ένωσης, της εγκαταστάσεις της Αφρικανικής Ένωσης αυτή η πρώτη διεθνής διάσκεψη για την ασφάλεια τροφίμων και θα περάσουμε και σε μια δεύτερη φάση αυτής της διάσκεψης που θα γίνει στη Γενέβη το Μάιο σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου για να δούμε πώς θα θεσπίσουμε κάποια κάποιες προδιαγραφές και συστάσεις για τα θέματα του εμπόριου. Έχουμε και ένα στόχο. Στο εμβληματικό μας πρόγραμμα στόχος μας είναι μέχρι το 2025 να τριπλασιάσουμε το ενδοαφρικανικό εμπόριο, τις ενδοαφρικανικές συναλλαγές. Και μάλιστα θα έχουμε την πρώτη διετή μας ε, έκθεση γιατί στο εμβληματικό μας αυτό πρόγραμμα ο έβδομος πυλώνας είναι η λογοδοσία, που συμφώνησαν και αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Όταν συνεργάζεται κανεί με εταίρου, θα πρέπει να λογοδοτεί, να παρακολουθεί την πρόοδο, να δίνει λογαριασμό. Και χώρε που ήταν πολύ ασθενεί ό,τι αφορά τον τριπλασιασμό του εδωαφρικανικού εμπορίου θα ενισχυθούν. Θα καταβάλουμε περισσότερε προσπάθειε για να βελτιώσουμε τον όγκο αυτού του εμπορίου. Και η επόμενη έκθεση που θα υποβάλουμε στους αρχικούς κρατών και κυβερνήσεων θα είναι το 2020. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τον απολογισμό για να δούμε πώς έχουν βελτιωθεί οι χώρες στις επιδόσεις τους. Σε ό,τι αφορά την Κίνα, αγαπητέ συνάδελφε, ε, νομίζω ότι η ερώτησή σας ε, αποτινόταν σε εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι τόσο στην Αφρικανική Ένωση, γιατί έχουμε αρκετέ εταιρικέ σχέσει με την Κίνα που λειτουργούν πολύ καλά. Φυσικά σεβόμαστε την κυριαρχία όλων των χωρών. Αλλά νο... άκουσα την ερώτησή σας ε, στα πορτογαλικά. Δεν ξέρω αν ε, δεν μεταφράστηκε σωστά αυτό που είπατε, αλλά νομίζω ότι η ερώτηση του κυρίου Σάντος ήταν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι προς την Αφρικανική Ένωση. μάλιστα. Ολοκληρώσαμε την πολύ σημαντική αυτή συζήτηση. Εδώ συνδυάσαμε την αφρικανική με την ευρωπαϊκή πείρα και εμπειρία για να βελτιώσουμε το ρόλο του αγροδιατροφικού κλάδου στη δημιουργία θέσεων απασχόληση, πιο βιώσιμο θέσεων απασχόληση και προ μια βιώσιμη ανάπτυξη και τη Αφρική. Πραγματικά αυτή είναι πολύ σημαντική πρόκληση. Πάντω το έργο και οι συστάσει τη ειδική ομάδα εργασία ε, στην οποία προέδρευσε ο κ. Άρνοντ θα μας βοηθήσουν να ενισχύσουμε τον αγροδιατροφικό κλάδο και είμαι βέβαια ότι θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό στην Επιτροπή, θα εγκύψουμε και πάλι σε αυτό το σημαντικό ζήτημα. Δεν έχω τίποτα άλλο παρά να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας, για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και πολύ ευχαρίστω θα σας υποδεχθούμε και στο μέλλον. Και δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστήσω θερμά τους παρόντες. Να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς, λέει η Πρόεδρος για την ανεκτήμητη, όπως πάντα, βοήθειά του στις συνεδριάσεις μας και να πω ότι διεκπαιρεώσαμε την ημερήσια διάταξη, εκτός αν, και έμεινε, αν έμεινε τίποτα για τα διάφορα. Αν δεν υπάρχει τίποτα στα διάφορα, ολοκληρώνεται η συζήτηση. Να σας υπενθυμίσω ότι η επόμενη μας συνεδρίαση θα γίνει στις 18 Μαρτίου. Σας ευχαριστώ και χαίρετε.